Se prendiamo posto cominciamo, grazie. Allora, l'approvazione, buongiorno a tutti. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ, εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη πρώτα απ' όλα. Σας έχει σταλεί το σχέδιο στις 7 ε, Νοεμβρίου ηλεκτρονικά. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι η συνεδρίαση αυτή ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο με εξαίρεση το τμήμα που έχει να κάνει με την ψηφοφορία για τον νέο διευθυντή της Όλαφ. Ξεκινάμε με το πιο σημαντικό θέμα στην σημερινή μας ημερήσια διάταξη που είναι η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2009. Θα μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κύριος Σίλβα Καλδέρα και χαιρετίζω εδώ την παρουσία του. Πριν όμως του δώσω το λόγο, θέλω να χαιρετήσω εδώ και τον πρόεδρο και τους ε, άλλους ε, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως επίσης και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκονται εδώ. Είναι η πιο σημαντική στιγμή στη δράση της Επιτροπής μας, γιατί έχουμε το προνόμιο εμείς να ακούσουμε για τη δουλειά ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας μιλήσει λοιπόν για τη χρήση των κολυδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και από τα κράτη-μέλη. Εγώ διάβασα την έκθεση αυτή με πάρα πολύ προσοχή και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά σημεία. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα τον Πρόεδρο. Πρόκειται λοιπόν για μια τεχνική δουλειά, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, και στη συνέχεια εμείς θα μπορέσουμε να εκφραστούμε, να πούμε την άποψή μας, να σκίσουμε τον δικό μας το ρόλο και να δούμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε να είναι αυτή όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και να διέπεται και από διαφάνεια. Θέλουμε να αποφύγουμε ανομαλίες όπως έχουν παρατηρηθεί πρόσφατα. Θέλουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους απάτη. Κύριε Καλέρα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, για μένα είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάσω σήμερα στην Επιτροπή σας την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την υλοποίηση του προϋπολογισμού και την ετήσια έκθεση για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2009. Έχει φτάσει η στιγμή για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η συνθήκη της Λισαβόνας ξεκίνησε τη διαδικασία το 2009. Το σχέδιο του νοσονομικού κανονισμού ε, καθορίζει ε, τις γενικές κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης και για φέτος, αλλά η επόμενη χρονιά θα είναι ε, καθοριστική για την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιάσω τα τέσσερα βασικά στοιχεία σε αυτή την ετήσια έκθεση και στη συνέχεια να υπενθυμίσω τα βασικά συμπεράσματα και συστάσεις των πρόσφατων γνωμοδοτήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν την μεγαλύτερη μεγαλύτερη σημασία για αυτή τη διαδικασία μεταρρύθμισης. Το, τα βασικά μηνύματα καλύπτουν την αξιοπιστία των λογαριασμών, την νομιμότητα και την κανονικότητα ε, των ε, πράξεων και μια σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτού του έτους με τα αποτελέσματα προηγουμένων ετών και τέλος ε, τις διορθώσεις λαθών επιπολιτού βάσεω. βάσεως. Καταρχήν, όσον αφορά τους λογαριασμούς, το ελεγκτικό συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν ε, σωστά τα οικονομικά αποτελέσματα και ε, τι χρηματοοικονομικέ ροε. Για τρίτο συνεχές έτος το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι δεν υπήρχαν ε, σφάλματα ε, στους λογαριασμούς και ότι είναι αξιόπιστοι. Η απουσία βέβαια ε, λαθών δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ασφαλμένων δηλώσεων στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη διαδικασία υποβολής των λογαριασμών, ιδίως όσον αφορά τους λογαριασμούς για προχρηματοδότηση συζήτηση ε, καθώς ε, και το διαχωρισμό των οικονομικών ετών, καθώς και το πώς λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις ε, δαπανών. Όσον αφορά την νομιμότητα και κανονικότητα, το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τα έσοδα δεν είχαν σημαντικά ασφάλματα και ότι ήταν αποτελεσματικά τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας. Όπως κατά τα προηγούμενα έτη, έτσι και φέτος οι δεσμεύσεις δεν είχαν σημαντικά σφάλματα και κάτι που πρέπει να τονίσουμε και φέτο είναι ότι οι πληρωμές που αφορούν τον προπολογισμό συνεχίζουν να έχουν σημαντικά σφάλματα εκτό από δύο τομεί δαπανών. Αυτέ οι δύο εξαιρέσει είναι οι διοικητικέ δαπάνε, όπου το σύστημα επί πολλά έτη ε, είναι ε, συνεπέ προ τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και ο άλλο τομέα είναι οι οικονομικέ και νομισματικές πολιτικέ. Σε όλου του άλλου τομεί, το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε σημαντικά σφάλματα. Στον τομέα τη γεωργία και των φυσικών πόρων, που αποτελούν περίπου το ίμιση του προπολογισμού, το ελεγκτικό συνέδριο εκτιμά το ποσοστό σφάλματος από 2 έως 5% είναι λίγο υψηλότερο από ό,τι κατά το περσινό έτος. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ε, συνάδει προς την αξιολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου και για τα δύο έτη ότι τα συστήματα αυτά είναι μόνο εν μέρη αποτελεσματικά. Τα περισσότερα σφάλματα προκύπτουν από την ε, υπερβολική δήλωση ε, επιφανειών που είναι επιλέξιμες για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και το καθεστώς ενιαίας θερματικής ενίσχυσης. Το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά να μειωθεί ο κίνδυνος φάλματος, βελτιώνοντας την ποιότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να διαπιστώνονται τα δικαιώματα και για να υπολογίζονται οι πληρωμές και ταυτόχρονα να διευκρινιστούν οι διατάξεις που ισχύουν για την χρησιμοποίηση και τη διατήρηση των γεών και οι ισχύουσες διατάξεις να εφαρμόζονται. Ο τομέα τη συνοχή είναι η δεύτερη ομάδα σημαντικών πολιτικών που αποτελεί σχεδόν το 1 τρίτο του προπολογισμού και εδώ είναι ο μόνο τομέα του προπολογισμού όπου το ποσοστό ε, εκτιμόμενου σφάλματο είναι πάνω από 5% και τα τρία τέταρτα των σφάλματων έχουν σχέση με σοβαρέ παραλήψεις εκ μέρου των εθνικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν σχέση με κρατικέ προμήθειε και τα υπόλοιπα αφορούν την πληρωμή μη επιλέξιμου κοστου μη επιλέξιμων δαπανών για σημαντικό τμήμα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από του δικαιούχου προ καταβολή των πληρωμών. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι περίπου το 1 τρίτο των σφαλμάτων που ανεβρέθησαν στι. Ε, ενδιάμεσε πληρωμέ και στι τελικέ πληρωμές θα μπορούσαν να έχουν ανοιχνευθεί και διορθωθεί από τα κράτη-μέλη πριν από την πιστοποίηση των δαπανών από την Επιτροπή. Έτσι έδειξαν τουλάχιστον οι έλεγχοι που έγιναν. Συνολικά, το Ελληνικό Συνέδριο αξιολογεί τα συστήματα στον τομέα τη συνοχή ε, ω εν μέρη μόνο αποτελεσματικά και έχει τέσσερι ε, συστάσει προ την Επιτροπή. Πρώτον, να ενθαρρύνει τι εθνικέ αρχέ να εφαρμόζουν αυστηρά του διορθωτικού μηχανισμού, πριν υποβάλουν τι δηλώσει δαπανών στην Επιτροπή. Δεύτερον, να διασφαλίσει ότι οι ανιχνευόμενες ε, μη επιλέξιμες δαπάνες δεν θα, αντικατα... θα αντικαθίστανται από τις εθνικές αρχές με άλλες δαπάνες που και αυτές θα είναι παράτυπες. Τρίτον, στο πλαίσιο του ρόλου της, της εποπτείας να φροντίζει για την σωστή λειτουργία των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου για την περίοδο 2007-2013. Και τέλος, να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις των κρατών μελών και την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές προμήθειες. Οι πληρωμές όσον αφορά την έρευνα τώρα, την ενέργεια και τις μεταφορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από το σφάλμα και τα συστήματα εξακολουθούν να είναι εν μέρη μόνο αποτελεσματικά. Όπω και το 2008, έτσι και τώρα το Λεκτικό Συνέδριο πιστεύει ότι το ποσοστό σφάλματο είναι ανάμεσα στο 2 και στο 5%. Τα σφάλματα αυτά έχουν να κάνουν με την αποζημίωση ε, κονδυλίων όσον αφορά δικαιούχους που έχουν ζητήσει χρήματα για προγράμματα στον τομέα της έρευνας. Όσον αφορά τώρα την ομάδα των πολιτικών που έχει να κάνει με την εξωτερική βοήθεια, την ανάπτυξη και την διεύρυνση, η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτή που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή υπάρχουν ε, πληρωμές που επηρεάζονται από ένα σημαντικό ποσοστό σφάλματος και έλεγχοι γίνονται μόνο εν μέρη. Το ποσοστό σφάλματος που εκτιμούμε είναι 2 με 5%. Τα σφάλματα αυτά έχουν να κάνουν με την επιλεξιμότητα των δαπανών, παρόλο που το ελεκτικό ε, συνέδριο έχει διαπιστώσει και πολλές περιπτώσεις όπου δεν τηρείται δεν τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέμα κρατικών προμηθειών και γι' αυτό και κάνει συστάσεις για βελτιωμένο έλεγχο των συστημάτων. Η εξωτερική βοήθεια χορηγείται από την Europe Aid στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Και δημοσιεύεται ξεχωριστή έκθεση για την βοήθεια αυτή κάθε χρόνο. Για το 2009 το Ελεκτικό Συνέδριο έχει εκφράσει γνωμοδότηση χωρίς επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των λογαριασμών, όμως πρέπει να ε, διαπιστώσουμε ότι τα συστήματα είναι εν μέρη μόνο αποτελεσματικά. Τα συστήματα ελέγχου όσον αφορά την κανονικότητα και την νομιμότητα των δαπανών. Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση και την ηθαγένεια, το Ελεκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε διάφορα ασφάλματα τα οποία έχουν να κάνουν με τέτοια προγράμματα για τις προηγούμενες προγραμματικές ε, περιόδους που έκλεισαν το 2009. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν στον τομέα της συνοχής. Και φτάνω στο τρίτο σημείο κλειδί της έκθεσής μας. Η εκτίμηση του σφάλματος για τη συνοχή ήταν χαμηλότερο από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές και για τον προπολογισμό στο σύνολό του το... ο μέσος όρος έχει πέσει σχετικά. Βέβαια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πριν καταλήξουμε σε συμπεράσματα όσον αφορά τις τάσεις που παρατηρούνται, γιατί υπάρχουν πολλές μεταβλητές όσον αφορά το είδος των πληρωμών που αλλάζει σε ένα μεγάλο βαθμό από τον ένα χρόνο στον άλλο. Για το 2009 έχουμε διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με το 2008. Παρ' όλα αυτά, η μείωση όσον αφορά το εκτιμούμενο ποσοστό σφάλματος για την συνοχή ήταν σημαντικό. Και έτσι αντισταθμίστηκε κάπως η αύξηση που είχαμε σε άλλους τομείς. Η εκτίμηση για το επίπεδο σφάλματος στο σύνολο είναι χαμηλότερο λοιπόν το 2009 σε σχέση με το 2008. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την τάση προς τα κάτω που αναφέραμε ήδη από πέρυσι. Όμως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Όπως είπα και νωρίτερα, τα συστήματα παραμένουν εν μέρη μόνο αποτελεσματικά για όλα τα είδη των πολιτικών μας, εκτός από τις διοικητικές δαπάνες. Συγχρόνως όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διαχείριση και έλεγχος είναι πολυετής. Σφάλματα λοιπόν στις πληρωμές που έγιναν το 2009 μπορεί να εντοπιστούν και να διορθωστούν τις επόμενες χρονιές χάρη στην λειτουργία του μηχανισμού πολιετών διορθώσεων. Έτσι λοιπόν το λεκτικό Συνέδριο και πάλι εξέτασε προσεκτικά τις πληροφορίες που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εισπράξεις και για άλλες οικονομικές διορθώσεις. Όμως η Επιτροπή διαπιστώνει και κάνει ε, πολλά θετικά βήματα το 2009 για να αυξήσει και να βελτιώσει τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με ε, τους λογαριασμούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πάντα αξιόπιστες γιατί σε τομείς όπως είναι η συνοχή για παράδειγμα υπάρχουν αδυναμίες των συστημάτων όσον αφορά την ενημέρωση για τις διορθώσεις αυτές που γίνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, οι περισσότερες διορθώσεις στις τιμές είναι δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη και αντιστοιχούν στην αδυναμία των διαφόρων συστημάτων. Αυτέ οι διορθώσει έχουν αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη να φροντίζουν να διορθώσουν τα συστήματά του και να προστατεύεται έτσι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, δεν επιτρέπει να διορθωθούν σφάλματα τα οποία εντοπίζονται από το ελεγκτικό συνέδριο ω επιτοπλίστων σχετικά με ποσά τα οποία δηλώθηκαν ε, λανθασμένα από τους δικαιούχους ή πληρώθηκαν λανθασμένα σε αυτούς. Το ελεκτικό συνέδριο λοιπόν συστήνει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν ε, τις πληροφορίες ε, και την κοινοποίηση που κάνουν σε σχέση με τα σφάλματα, ώστε οι πληροφορίες που έχουμε να είναι σωστές και να λαμβάνονται σωστά υπόψη στους λογαριασμούς για τον μηχανισμό πολιετών διορθώσεων. Έτσι φτάνω εδώ στο τελευταίο μήνυμα κλειδί που περιλαμβάνει η έκθεσή μα, που είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών ε, που δίνει όσον αφορά την ίσπραξη των ε, αδίκως ε, πληρωμένων ποσών. Όμως οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πει ότι μπορούν να συγκριθούν σωστά ειδικέ πληροφορίε με τι διορθώσει που δίνει το ελεγκτικό συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Πρέπει να αναλάβουμε διάφορες πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την οικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει ένα σχέδιο για την επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιαστεί μέσα στα 2011 και θα είναι ένα σχέδιο κανονισμού που θα καθορίζει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα σχέδιο απόφασης σε σχέση με τους ίδιους πόρους και τις νομοθετικές προτάσεις που γίνονται για να τεθούν σε εφαρμογή πολιτικές και προγράμματα που έχουν να κάνουν με τους κύριους τομείς δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Το κύριο πάντως μήνυμα του Λεκτικού Συνεδρίου είναι να αντιμετωπιστούν οι κύριε πηγές κινδύνου όσον αφορά την διαχείριση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ό,τι είπαμε ήδη στην αρχή της χρονιάς που είχαμε εκδώσει την γνωμοδότησή μας ισχύει. Ότι δηλαδή πρώτα απ' όλα το ποσοστό σφάλματος εξακολουθεί να είναι υψηλό σε διάφορους τομείς του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη συνοχή. Δεύτερον, τα ασφάλματα τα οποία εντοπίζονται από το ελεκτικό συνέδριο απορρέουν κυρίως από λάθος πληρωμές που έχουν γίνει σε δικαιούχους ή από λάθος αιτήσει που έχουν γίνει από τους δικαιούχους, κυρίως στον τομέα των κρατικών προθυμηθειών. Τρίτον, υπάρχουν δύο τρόποι για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Είτε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα διαχείριση, ιδίω με μηχανισμού ίσπραξη και με διορθώσει πιο αποτελεσματικέ, ή να απλοποιήσουμε του κανόνε και του κανονισμού. Τέταρτον, το ελεγκτικό συνέδριο εντοπίζει διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται ξανά και ξανά στις ειδικέ εκθέσεις και έχουν να κάνουν με διάφορα προγράμματα δαπανών. Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση προτείνουμε να εφαρμοστεί ένα σύνολο αρχών όταν επανεξετάζονται τα προγράμματα δαπανών θέτοντας τα εξή ερωτήματα. Τα προγράμματα είναι μια επιπλέον αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν κάποια προσθέμενη αξία. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι και το καθεστώς δαπανών είναι ε, αποτελεσματικό, είναι ρεαλιστικό. Το καθεστώς είναι αρκετά απλό και η υποχρέωση να ε, επιστρέφονται οι λογαριασμοί είναι κάτι το οποίο αναφέρεται ξεκάθαρα. Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση της ποιότητας των δαπανών. Αυτό πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Και η απλοποίηση των νομοθετικών πλαισίων και η δημιουργία συστημάτων ελέγχου πιο αποτελεσματικών για να, για να μειωθεί το ποσοστό και ο κίνδυνος σφάλματος. Έτσι θα βελτιώσουμε ε, την κατάσταση και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Χρειάζεται απλοποίηση επίσης της νομοθεσίας ανατομέα. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μόνο αν έχουμε προτάσεις για νομοθεσία ανατομέα ε, έχει νόημα και σύστασή μας. Και αυτό γιατί έτσι εντοπίζονται οι κανόνες νομιμότητας και κανονικότητας για τους λογαριασμούς, αλλά βελτιώνεται και ο έλεγχος και η διαχείριση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται και που είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων δαπανώνται σωστά και αποτελεσματικά και υπεύθυνα από όλου μα. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν προτείνει νομοθεσία και φροντίζει για την χρήση των κονδυλίων αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Τα κράτη-μέλη επίσης στα πλαίσια της δικιάς τους καθημερινής διαχείρισης για περίπου 80% του προπολογισμού. Επίσης και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που είναι συνομοθέτες έχουν τη δικιά τους ευθύνη στην νομοθετική διαδικασία και βέβαια τέλος το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο αποτελεί και τον εξωτερικό ελεγκτή για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελεγκτικό συνέδριο σκοπεύει να αναλάβει πλήρω τις ευθύνες του ώστε να διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια διαπανώνται ορθά, καλά και αυτό το κάνει με την ε, δημοσίευση των ετησίων εκθέσεών του για την εκμετάλλευση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά εσάς κύριε Πρόεδρε, κύριε Καλντέρα και κατά αυτόν τον τρόπο ε, ανοίγουμε το έργο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού που θα οδηγήσει ε, στη συνέχεια στην απαλλαγή. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη, θα ήθελα να δώσω καταρχήν το λόγο στην Επιτροπή. Αγαπητέ Πρόεδρε Καλτέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαπόλτζο, αξιότιμα μέλη αυτής της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι απαντήσεις της Επιτροπής προκύπτουν από τον επικοδομητικό διάλογο μεταξύ Επιτροπής και Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Καλτέρα και τα μέλη της Επιτροπής για την εξαιρετική συνεργασία. Η ετήσια έκθεση της έκθεσης περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο μία ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιδόσεων, αλλά και πολύτιμες πληροφορίες επί των οποίων θα, η Επιτροπή θα συναγάγει ε, συμπεράσματα για να καθορίσει τις νέες πολιτικές και τον νέο προϋπολογισμό. Χαίρομαι το, ε, που το ελεκτικό συνέδριο διαπιστώνει ε, πρόοδο στον αντικειμενικό τρόπο παρουσίασης ε, των θεμάτων. Διαπιστώνουμε επίσης κάποια κριτική και αποτελεί δέσμευση της Κομισιόν αλλά και μου προσωπικός να καλύψουμε αυτά τα κενά τα οποία επισημαίνονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να απαντήσω στα βασικά μηνύματα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου που αποτελούν και βάση ε, για την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Καταρχήν, οι ετήσιοι λογαριασμοί σε ε, τρίτη ε, συνεχή χρονιά δέχονται μια θετική γνωμοδότηση χωρίς επιφυλάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα διότι τούτο επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων των ε, λογιστικό μας ε, συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις ε, διορθώσεις όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή σας μετά από τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Ελεκτικό Συνέδριο επισημαίνει επίσης κάποιες αδυναμίες. Η, ως προς την άμεση καταγραφή των λογαριασμών και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Τούτο όμως ε, δεν οδηγεί σε ε, επιφυλάξεις. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να βελτιώνει τις καθημερινές της πρακτικές τήρησης των λογαριασμών. Ως προς το θέμα αυτό θα ήθελα να επισημάνω επίσης τα βασικές τιμές και στοιχεία των τυσίων ε, λογαριασμών για το 2009. Υπήρξε ένα πλεόνασμα 2,26 δις ευρώ, ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος που οφείλεται στην εφαρμογή των δαπανών σε κάποιους τομείς και τα πιο σημαντικά ήταν ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ως προς τον ισολογισμό βλέπουμε μια αύξηση των δανείων 7,2 δις ευρώ ε, που οφείλονται ακριβώς σε δάνεια που χορηγήθηκαν το 2009 τούτα θα περιληφθούν ε, στα οικονομικά αποτελέσματα των, ε, του ενεργητικού. Η αύξηση της χρηματοδότησης αυξήθηκε κατά 9,5 δις ευρώ. Ιδιαίτερα ως προς το τρίτο σκέλος των, της πληρωμής διαρθωτικών ταμείων 2007-2013. συνολική χρηματοδότηση είναι 47,8 δις ευρώ. Ως προς το παθητικό έχουμε μία μείωση κατά 7,2 διότι ε, έγινε μία μείωση ως προς τις ε, ε, ετήσιες αυξήσεις του προσωπικού. Ως προς την νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών, χαίρομαι για την θετική γνώμη του ελεγκτικού συνεδρίου και έχει μειωθεί ο αριθμός των φαλμάτων το 2009, όπως είπε ο πρόεδρος Καρδέρα νωρίτερα. Ε, ε, υποχρεώσεις για τον συνολικό προϋπολογισμό και τις ε, εκκρεμείς δαπάνες είναι ελεύθερες από οποιοδήποτε σφάλμα. Και εδώ υπάρχει μια θετική τάση για τη μείωση των σφαλμάτων όπως επισημώνεται από το ελεκτικό συνέδριο στους τομείς ενέργειας και μεταφορών. Στον τομέα της γεωργίας ε, το ποσοστό σφάλματος είναι γύρω στο 2%. Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται από το συνέδριο είναι γνωστοί και αντιμετωπίζονται από την Κομισιόν καλύπτονται επαρκώς από την ειδική διαδικασία συμμόρφωσης που έχει σχεδιαστεί για ώστε να εξαιρούνται οι δαπάνες οι οποίες ε, δεν γίνονται από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, την περασμένη Παρασκευή η Κομισιόν αποφάσισε να ζητήσει πίσω ένα σύνολο 105 δις από τις χώρες μέλη για ποσά τα οποία δεν δαπανήθηκαν ορθώς από τις χώρες μέλη. Τώρα, ως προς τους άλλους τομείς πολιτικής. Το ποσοστό σφαλμάτων για την παιδεία και τον πολιτισμό είναι γύρω στο 2% και έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την εξωτερική βοήθεια, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση, όπου το ποσοστό σφάλματος παραμένει μεταξύ 2 και 5%. Για πρώτη φορά στα χρονικά το συνέδριο υπολογίζει ότι συνολικά το ποσοστό σφάλματος είναι γύρω στο 2 με 5%. Τούτο σημαίνει ότι πάνω από το 95% των πληρωμών είναι ε, ελεύθερες από σφάλματα. Είναι ένα θετικό δείγμα ε, και αποδεικνύει ότι οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη στις ουσιαστικές μειώσεις του το, σφάλματο, το ποσοστού σφάλματος στην συνοχή, στον τομέα της συνοχής. Έχουμε δηλαδή μια πιο προσεκτική προσέγγιση και το τούτο θα επεκταθεί και στους τομείς όπου έχουν εντοπιστεί σφάλματα. Είναι επίσης αποτέλεσμα ε, και της ε, διαδικασίας αξιολόγησης ε, της συμμόρφωσης και της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρών μελών και των συστημάτων που αξιολογούνται διαρκώς. Ωστόσο, συμμερίζομαι την άποψη του Προέδρου Καλντέρα για τον περιορισμό των σφαλμάτων στον τομέα της συνοχής. Το νέο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης 2007-2013 ε, είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τους προηγούμενους ελέγχους εντοπισμού ε, σφαλμάτων και λαθών. Την έκθεσή του το Ελεκτικό Συνέδριο τονίζει την ε, ανάγκη να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία ώστε να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα και επισημαίνει τη σημασία των, της ορθής πληροφόρησης. Αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Η αύξηση του ύψους των κονδυλίων όπου εντοπίζονται σφάλματα από πλευράς εθνικών χωρών ε, είναι κάτι που επισημαίνεται οι διορθώσεις που εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν το 2009 ανέρχονται σε 3,3 δις ευρώ. Επισημαίνεται ακόμα η ε, υπάρχουσα αδυναμία σε κάποιους τομείς τουλάχιστον από πλευράς εθνικών χωρών στην υποβολή των πληροφοριών τους. Ε, κατά την άποψή μου ο σχεδιασμός πιο αποτελεσματικών μηχανισμών, απλοποίηση των κανόνων επιλεξιμότητας που θα αποκλείουν τα σφάλματα και η βελτίωση της ε, ποιότητας και της αξιοπιστίας ε, των πληροφοριών που έρχονται από τις χώρες μέλη θα οδηγήσουν στην βελτίωση. Αυτό είναι μόνο ένα στοιχείο της ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σύμφωνα με τις νέες διατάξεις προβλέπεται από το άρθρο 317 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά τούτο δεν είναι αρκετό. Πεποίθησής μου είναι ότι οι ε, δημοσιονομικοί παράγοντες θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια ώστε να υπάρξει ποιοτική ε, βελτίωση των δαπανών. Ε, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας και ε, κατά κύριο λόγο εξαρτάται το αποτέλεσμα από την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας. Απαιτείται λοιπόν καθορισμός σαφών και μετρήσιμων στόχων και συστημάτων που θα παρακολουθούν την πρόοδο και τις επιπτώσεις των ενεργειών μας. Αξιότιμα μέλη αυτής της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, πρέπει να ε, συνεχίσουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα, να καλύψουμε τις αδυναμίες που επισημαίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσω και το σχέδιο για την απαλλογή ε, για το 2009-2010. Περιλαμβάνει τις βασικές στρατηγικές και τα βήματα που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε ε, μια θετική εξέλιξη. Υπό το φως της ετήσιας έκθεσης του 2009 μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτή η ατζέντα παραμένει σχετική για τις μετονικές μας ενέργειες. Τελειώνοντας, με χαρά επισημαίνω ότι η έκθεση του 2009 έχει θετικά αποτελέσματα. Συνιστά ένα ε, σημαντικό και έγκαιρο στοιχείο προς την κατεύθυνση πιο αποτελεσματικής δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας οδηγήσει στις επόμενες γενναίες προγραμμάτων. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ο κύριο Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική παρουσίαση που μας κάνατε στην Επιτροπή μας. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια θετική τάση όσον αφορά ε, τη διατύπωση των ασφαλμάτων και ο κ. Σέμετε πολύ σωστά ε, είπε αυτό που ε, είχε, είχε ξεκινήσει ο κ. Σιμ Κάρλας ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Είναι θετική αυτή η τάση όσον αφορά τη διατύπωση των ασφαλμάτων και πρέπει να το επισημάνουμε. Υπάρχει σημαντική βελτίωση στον τομέα της συνοχής σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ένα από τα βασικά ε, ε, ε, κομμάτια των δαπανών του προϋπολογισμού και πρέπει να δούμε και τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν στον τομέα της γεωργίας. Η συνοχή είναι μια πολιτική που αφορά χώρες που χρειάζονται τη βοήθεια αυτή. Οι χώρες που έχουν επιλεγεί συνήθως είναι μικρές χώρες και πολύ συχνά ανήκαν στην ε, Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Εδώ στατιστικά έχουμε μια θετική εξέλιξη. Συμφωνώ με την εκτίμηση του Προέδρου και το ανέφερε αυτό και η Επιτροπή ότι τα στοιχεία παρουσιάζουν διακύμανση και δεν πρέπει να ε, υπερβάλλουμε στην αξιολόγησή μας και θα πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να μην υπερβάλλουμε και όσον αφορά την επιδείνωση των σφαλμάτων στον τομέα της γεωργίας. Ε, παρατηρούμε τις μικρές διακυμάνσεις που υπάρχουν και τις λαμβάνουμε υπόψη μας και ενδεχομένως ε, μέσω ενός διαλόγου μεταξύ Επιτροπής και Ελεκτικού Συνεδρίου να μπορούν αυτές οι λεπτομέρειες να ληφθούν υπόψη καλύτερα χωρίς να υπερβάλλουμε στην αξιολόγηση αυτών των μικρών διακυμάνσεων. Πρέπει όμως να διαπιστώσουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στου τομεί αυτούς όπου διαπιστώνονται τα σφάλματα. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή, και μιλάμε για το 80% των δαπανών που είναι σε από κοινού διαχείριση ε, υπάρχουν τεράστια προβλήματα και διαπιστώνουμε ότι σε πολλούς τομείς υπάρχουν πηγές σφάλματος και η Επιτροπή δεν καταλήγει πάντοτε σε κυρώσεις. Στο παρελθόν η Επιτροπή διαπίστωνε σφάλματα, διαπίστωνε τομείς όπου υπήρχαν έργα που δεν ήταν ε, σωστά, αλλά συνέχισε να τα χρηματοδοτεί για πολιτικούς λόγους. Παρότι ε, ήδη από το 2005 είχε μέτρα για επιβολή κυρώσεων, όπως παραδείγματο χάρη στον τομέα της γεωργίας με το άρθρο 17 του κανονισμού 1290 θα μπορούσε η Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές αμέσως μόλις διαπίστωνε σφάλματα και για συγκεκριμένο κράτος μέλος ε, για την Ελλάδα, ένα από τα παλιά κράτη-μέλη, επί 10 χρόνια στον τομέα της γεωργίας δίδονταν σφάλματα, δίδονταν συγγνώμη δαπάνες, παρότι δεν είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα επιτήρησης και ελέγχου που θα έπρεπε να έχουν ε, χρησιμοποιηθεί. Και το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας. Υπάρχει λοιπόν το εύλογο ερώτημα γιατί ο φορολογούμενος, τον οποίο εκπροσωπούμε εμείς εδώ, ε, γιατί οδηγείται σε αυτή την κατάσταση όταν υπάρχουν ε, σφάλματα και ανέφερα μόνο ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Όταν υπάρχουν σφάλματα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε κυρώσεις. Έχουμε τα νομικά μέσα στη διάθεσή μας και πρέπει να εφαρμόσουμε τις κυρώσεις αυτές. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κράτη-μέλη στα οποία έχουν διαπιστωθεί τα σφάλματα που μας αναφέρετε στην έκθεσή σας. Έχουμε όμως ε, τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εδώ σε αυτό το τεύχος που είναι πολύ ενδιαφέρον και στην σελίδα 111 μπορείτε να δείτε τους ε, μεγαλύτερους παραπτωματίες <laughs> θα λέγαμε και υπάρχουν χώρες που ήδη από το 2009 θα έπρεπε να πληρώσουν περισσότερα και θα θέλω να τις αναφέρω είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τέσσερις χώρες που θα έπρεπε να πληρώσουν, να επιστρέψουν χρήματα. Λοιπόν, τι συμβαίνει κυρίες και κύριοι όταν κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τι κάνει η Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση και τι κάνουμε κι εμείς. Οι πηγές φαλμάτων υπάρχουν, είναι γνωστέ εδώ και χρόνια, αλλά δεν ακολουθεί πάντοτε την απαιτούμενη διαδικασία η Επιτροπή. Όταν διαπιστώνεται ένα σφάλμα, θα πρέπει να ισχύει ο κανόνα του 50-50. Θα πρέπει ε, ο, αυτός που διαπράττει το σφάλμα να πληρώνει το 50% ενώ τελικά πληρώνει μόνο το 10% και τελικά τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο εθνικό προπολογισμό, Άρα ο φορολογούμενο επιβαίνεται ει διπλούν. Έχει γίνει μια εσφαλμένη πληρωμή και στη συνέχεια υπάρχει μια κύρωση που επιβαρύνει τον εθνικό προπολογισμό και όχι το δικαιούχο ο οποίο ήταν η αιτία του σφάλματο, Δεν είναι αποδεκτό λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει μια γενική τάση λοιπόν θετική, αλλά σε ε, ε, επιμέρους περιπτώσεις υπάρχουν σφάλματα τα οποία πρέπει ε, να προσέξουμε και να διορθώσουμε και συμβαίνουν σφάλματα ε, όχι μόνο εκεί όπου έχουν κοινή διαχείριση η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και πολλές φορές ε, ε, λέμε ότι τα κράτη-μέλη φταίνε και όχι η Επιτροπή. Η συνθήκη όμως αναφέρει σαφώς ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κανονικότητα όλων των πληρωμών, ακόμη και για την περίπτωση που έχουν διαπράξει σφάλματα τα κράτη-μέλη και χειρότερες είναι, χειρότερα είναι τα σφάλματα στα οποία η Επιτροπή και μόνη είναι υπεύθυνη. Και θα ήθελα να αναφέρω ε, ένα παράδειγμα και νομίζω το ανέφερε και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το πρόγραμμα σχετικά με την εκπαίδευση όταν ε, το 24% της δειγματοληψίας, το 1 τέταρτο δηλαδή, διαπιστώνει σφάλματα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ε, τότε διαρωτώμε γιατί δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, γιατί μιλάμε για πόρους που διατίθενται απευθείας από την Επιτροπή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι το 1 τέταρτο του δείγματο ε, παρουσιάζει σφάλματα, αξίζει τον κόπο να διαρωτηθούμε γιατί υπάρχουν τόσα σφάλματα. Τώρα που έχουμε λάβει την ε, έκθεση θα μπορούσαμε ίσως να καλέσουμε και την Επίτροπο την κυρία Βασιλείου που είναι τώρα υπεύθυνη, δεν ήταν πριν υπεύθυνη για αυτά τα προγράμματα, αλλά είναι τώρα υπεύθυνη για αυτά τα προγράμματα και θα μπορούσε να μας απαντήσει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ε, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση που έχουμε άμεση σχέση Επιτροπής και πολιτών. Το ίδιο και στον ευρύ τομέα της έρευνας και καινοτομίας και εκεί υπάρχουν έργα τα οποία έχουν πολλά ασφάλματα. Περνάω στην ε, ευθύνη της Επιτροπής τώρα. Ανέφερα την συνθήκη ήδη και διαρωτώ με γιατί, όπως και πριν, η Επιτροπή δεν παρουσιάζει τη συνθετική έκθεση για τις δραστηριότητες. Γιατί δεν υπογράφει αυτή την έκθεση. Μέχρι τώρα υπογράφουν οι γενικοί διευθυντές την έκθεση αυτή και θα ήθελα να διεξαχθεί μια σχετική συζήτηση. Ο αρμόδιος επίτροπος ε, που έχει την πολιτική ευθύνη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αυτή. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής ή ο κύριος Σέμετερ, υπεύθυνο επίτροπος ε, για τα θέματα ελέγχου και κανονικότητες. Ε, πάντως κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Μέχρι τώρα και σε επίπεδο κράτους μέλους και Υπουργοί Οικονομικών πώς μπορούν να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτά τα οποία έχουν ε, κάνει οι διοικήσεις τους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτά τα οποία είναι στην αρμοδιότητά μας ε, να είναι και μέσα στον τομέα ευθύνης μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, γιατί αυτό είναι στοιχείο μιας δημοκρατίας αν ε, δεν ε, έχετε εμπιστοσύνη στο σύστημα ελέγχου και επιτήρησης και γι' αυτό δεν υπογράφετε, ε, τότε πρέπει να βελτιωθεί αυτό το σύστημα ελέγχου και επιτήρησης και πολύ σωστά το παρατηρεί το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του και το βλέπουμε στη συνοπτική έκθεση ότι υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα στο σύστημα ελέγχου. Δεν λειτουργεί δηλαδή το σύστημα ελέγχου όπως θα θέλαμε και δεν είναι αποδεκτό αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λειτουργεί και ευχαριστούμε τη συνάδελφο κυρία Γκρέσλε που μίλησε την περασμένη φορά στο Στρασβούργο για ένα σύστημα ελέγχου και επιτήρησης και για το πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα όταν γίνονται σωστά. Και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκρέσλι για αυτή τη, τη συνεισφορά. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στο μέλλον. Το συζητάμε αρκετό καιρό, μιλάμε για την κανονικότητα και λέμε ότι η νομιμότητα και η κανονικότητα είναι ένα βασικό θέμα. Και το θέμα της ε, νομιμότητας και της ε, κανονικότητας ε, άπτεται και της αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είναι αποτελεσματική και αποδοτική η Επιτροπή. Είναι πολιτικό τη στόχος αυτός. Και γι' αυτό χρειάζεται ανάληψη ευθυνών. Πρέπει να υπάρχουν έναντι των φορολογουμένων. Την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα πρέπει να έχουμε τρόπο να την αξιολογήσουμε. Μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε ένα νέο μέσο, της εκθέσεις αξιολόγησης που θα πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή στο μέλλον, αλλά αυτό είναι κάτι καινούριο. Ε, το συζητήσαμε εν ολίγης ε, με ε, τον Επίτροπο, με τον κύριο Σέμετα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τα KPIs, τα Key Performance Indicators, βασικοί δείκτες απόδοσης που θα πρέπει για κάθε πρόγραμμα να καταρτίζονται. για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να έχουμε ε, στοιχεία για το αν έχει επιτύχει το πρόγραμμα τον πολιτικό του στόχο. Γιατί περί αυτού πρόκειται, περί πολιτικών στόχων τους οποίους έχουμε συμφωνήσει και τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε. Και γι' αυτό θέλουμε και αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης. Μαζί με τη συνθετική έκθεση θα θέλαμε να έχουμε και μια έκθεση που να μιλά για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Και περνώ στο τελευταίο σημείο θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της απαλλαγής. Είναι μια συνήθις διαδικασία. Είναι πολύ νωρί ακόμη να μιλήσουμε για το αν θα δοθεί απαλλαγή ή όχι. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε τώρα είναι το ε, θέμα του αν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ε, διαδικασία προϋπολογισμού, αν χρειαζόμαστε περισσότερο τον προϋπολογισμό. Βλέπουμε και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που διαπιστώνει ότι για άλλη μια φορά υπάρχουν πολλά σφάλματα στη διαχείριση της Επιτροπής και σημαντικά όπως είπα σε πολλές ε, περιπτώσεις. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν θα πρέπει να δίδονται περισσότερα χρήματα σε αυτή την Επιτροπή. Γιατί να μην χρησιμοποιεί τα χρήματα που έχει ήδη διαθέσιμα βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολύ υψηλά ποσά τα οποία πρέπει να ανακτήσει η Επιτροπή, πρέπει να επιστρέψουν οι δικαιούχοι, τεράστια χρηματικά ποσά. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσει η Επιτροπή αυτά τα ήδη διαθέσιμα χρήματα. Και στη σελίδα 12 είναι η πιο σημαντική πρόταση της έκθεσης πιστεύω. Η έκθεση λέει στη σελίδα 12 ότι κατά την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου υπάρχουν σημαντικά ασφάλματα και τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας μόνο εν μέρη είναι αποτελεσματικά. Αυτή είναι η κεντρική πρόταση της έκθεσης, αυτή την πρόταση πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και αυτή την πρόταση πρέπει να προχωρήσουμε σε συζητήσεις με την Επιτροπή γιατί θα ζητούνται περισσότερα χρήματα και περισσότεροι πόροι πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί για έκτη φορά να διαπιστώνουμε σφάλματα και να μην κάνουμε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ ε, τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνεδρίου για τα θέματα τα οποία ανέφερε. Αναφέρατε τέσσερι συστάσει προ τι οποίε πρέπει να κινηθούμε και σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Γιατί πρέπει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να έχει προστιθέμενη αξία και αυτό πρέπει να καταδεικνύεται. Και είναι σημαντικά αυτά τα τέσσερα ε, θέματα, οι τέσσερι ερωτήσει και συστάσει που αναφέρετε. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη μελλοντική μα συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε την συζήτηση τώρα με τους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Μπάλστης πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού του Δουλεκτικού Συνεδρίου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο που ήρθε και μας παρουσίασε μια τόσο πλήρη έκθεση. Πρέπει επίσης να πω ότι συγκρίνοντας με το 2008 η τρέχουσα έκθεση για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι έχει μειωθεί το ποσοστό. Εμένα πάντως με ανησυχεί κάπως η παρουσίαση του λεκτικού συνεδρίου που λέει ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την ίσπραξη οφειλόμενων ποσών, οι πληροφορίες οι σχετικές δεν είναι αξιόπιστες. Και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Χατζημαρκάκη, για το ότι υπάρχουν προβλήματα που διαπιστώνονται και παρατηρούνται ξανά και ξανά κάθε χρόνο ακριβώς επειδή υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και αυτό είναι ένας τομέας πάνω στον οποίο πρέπει να δουλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για το 2009. Το 2009 εξετάσουμε τις δαπάνες των ε, προηγούμενων ε, περιόδων. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο να δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να βελτιώσει τη δουλειά της. Υπάρχει γεωργία, υπάρχει η συνοχή που αναφέρθηκε και νωρίτερα, Αυτοί είναι δύο τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Επίτα, τα οικονομικά και δημοσιονομικά επίσης είναι ένα σημαντικό τομέας. Εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν και βλέπουμε εδώ ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σφάλματος. Μιλάμε επίσης για την επιλεξιμότητα. 62% εκρατικές προμήθειες, παραβίαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτοί είναι τομεί στους οποίους παρατηρείται υψηλό ποσοστό σφάλματος. Τα κράτη-μέλη λοιπόν, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και τρεις μιλάμε επίσης για προβλήματα στις κρατικές προμήθειες, άρα επιβάλλεται μια σημαντική αλλαγή. Ίσως να λείπει η πολιτική βούληση κάποιων κρατών μελών και γι' αυτό και ρωτώ τον αρμόδιο επίτροπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι βήματα προβλέπει να κάνει προκειμένου να βελτιώσει το θέμα των κρατικών προμηθειών, να βελτιώσει το σύστημα ελέγχων και κυρίως την ε, διαχείριση των ελέγχων των πληρωμών. Πότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα η κοινωνία των πολιτών θα έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες που πρέπει να δίνουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. το τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον πρόεδρο του Λεκτικού Συνεδρίου για αυτά που μας είπε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα. Θα μπορούσαμε να καθίσουμε με ώρες να συζητάμε και να φιλοσοφούμε αν κάτι είναι καλό, αν είναι κακό, αν είναι μια πρόοδος, η οπισθοχώρηση. Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από το σημείο κίνησης και εξαρτάται επίσης και από τους στόχους που βάζουμε, τις προσδοκίες μας. Όταν μιλάμε για τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση είναι καταστροφική εδώ και πολλά χρόνια και το έχουμε ήδη πει αυτό. Ως εκπρόσωπος λοιπόν των φορολογούμενων και όλοι εμείς εκπρόσωποι των φορολογούμενων έχουμε υψηλές προσδοκίες σε όλους τους τομείς. Κάθε χρόνο περιμένουμε να δούμε πρόοδους σε όλους τους τομείς. Σε ορισμένους τομείς όντως υπάρχει πρόοδος και αυτό μας χαροποιεί. Είναι θετικά, για παράδειγμα, τα πράγματα όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής ή τα Διορθωτικά Ταμεία. Σε άλλους τομείς όμως υπάρχουν οπισθοχωρήσεις, όπως είναι η γεωργία, όπως είναι η φυσική πόρη. Συμφωνώ απόλυτα για το ότι δεν πρόκειται για πολύ μεγάλα ποσά, αλλά εμείς περιμένουμε πρόοδους σε όλους τους τομείς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σημείο κίνησης από το οποίο ξεκινήσαμε ήταν πολύ κακό. Έχω λοιπόν να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ίσως να μην έχω διαβάσει τα πάντα ε, και γι' αυτό ρωτάω όλα. συγκρίνουμε την ετήσια έκθεση του 2008 με την έκθεση που έχουμε στα χέρια μας και εδώ θα σας πω στα αγγλικά τι λέει το κείμενο, μας λέτε ότι το ελεγκτικό συνέδριο έκανε μια δειγματοληπτική έρευνα βάσει της οποίας λέει ότι ορισμένα ποσά δεν αποζημιώθηκαν. Και εγώ δεν τα βρίσκω τα ποσά αυτά στην ε, έκθεσή σας. Θέλω λοιπόν να ξέρω γιατί δεν αναφέρονται αυτά στην έκθεση που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Θέλω επίσης να αναφερθώ περισσότερο στον όρο σφάλμα. Όταν μιλάμε για σφάλμα, τουλάχιστον στη δικιά μου γλώσσα στα δανέζικα, μπορεί να σημαίνει κάτι όχι πολύ σημαντικό. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν κάποιο σφάλμα, όλοι κάνουν σφάλματα. Δεν είναι όλα τα σφάλματα σοβαρά. Το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του μας λέει ότι από τη στιγμή όπου πρόκειται για απάτη, τότε σημαίνει ότι από πρόθεση χρησιμοποιήθηκαν στραβά τα κοινοτικά κονδύλια. Εγώ δέχομαι το δικό σας τον ορισμό, αλλά θέλω να ξέρω σε πόσες περιπτώσεις υπήρξε πραγματικά πρόθεση. Με τα παραδείγματα που μας δώσατε εσείς, αν κοιτάξουμε τη σελίδα 9, στα δανέζικα τουλάχιστον, που μιλάμε για τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους, λέτε ότι διαπιστώνουμε πως όλες οι χώρες μέλη συστηματικά υπολογίζουν λανθασμένα τις επιφάνειες. Λέτε ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα εδώ με τις πληρωμές. Λέτε δηλαδή ότι συστηματικά τα κράτη-μέλη κοινοποιούν λανθασμένα δεδομένα. Εδώ πρόκειται για ένα λάθος ή πρόκειται για μια απάτη ηθελημένα. Αν πάρετε ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Για το Ταμείο Συνοχής, σελίδα 12 στα δανέζικα πάντα. Υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα εδώ που λέει ότι έχετε κάποια προβλήματα όσον αφορά συμβάσεις και ότι μερικές φορές πληρώσαμε έργα τα οποία δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. Εδώ πάλι πρόκειται για ένα λάθος ή πρόκειται για μία απάτη, για κάτι που έγινε από πρόθεση. Τα πράγματα, θέλω να πω, δεν είναι πάντα εύκολο να τα καταλάβει κανείς έτσι όπως διατυπώνονται δεν καταλαβαίνω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ενώ το σημαντικό είναι να ξέρουμε κατά πόσο πρόκειται για ένα λάθος που κατά λάθος έγινε ή αν πρόκειται για μια πρόθεση που υπάρχει από πίσω. Αν διαβάσετε λοιπόν ε, ένας άνθρωπος διαβάσει την έκθεση του λεκτικού συνεδρίου δεν καταλαβαίνει πότε υπάρχει πρόθεση και πότε όχι. Στη Γεωργία φαίνεται ότι έχουν γίνει μεγάλα λάθη. Εσείς έχετε παραδείγματα για τομείς όπου δεν έχουν γίνει. Κάθε φορά που διαπιστώνουμε ένα λάθος είναι για να υπάρξει κάποιο κέρδος. Στη σελίδα 32 επίσης το ελεγκτικό συνέδριο μας λέει ότι υπάρχουν μόνο τρεις περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να παρέμβει η Όλαφ για περιπτώσεις απάτης. Τρεις περιπτώσεις ετησίως. Και στα δύο παραδείγματα που αναφέρθηκαν όπου συστηματικά τα κράτη-μέλη δίνουν εσφαλμένες πληροφορίες και ξέρετε ότι ορισμένοι άνθρωποι πληρώθηκαν για πράγματα για τα οποία δεν αναφέρει τίποτα η σύμβαση, τι περιπτώσεις είναι αυτές, δεν θα πρέπει η Όλαφ να έχει παρέμβει. Όταν αναφέρετε λοιπόν συγκεκριμένα παραδείγματα, εγώ θέλω να μου πείτε γιατί δεν αναφέρετε, δεν κατονομάζετε τις χώρες οι οποίες έκαναν τα σφάλματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τη συνεργασία σας και τη βοήθειά σας κατά άλλα. Ο κύριος Ανδρέας τώρα έχει το λόγο. Η κυρία Ανδρέα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση. Κύριε Καλτέρα, λέτε ότι η βελτίωση στα ταμεία συνοχής ε, είναι σημαντική και είναι μεγαλύτερη αυτής ως προς τα γεωργικά. Τούτο αφορά τα συστήματα ελέγχου της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι συνολικά τα συστήματα απέτυχαν, άρα πρέπει να αρχίσουμε εκ του μηδενός. Θεωρείται ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε θετική τροχιά ως προς την νομιμότητα και την κανονικότητα. Αναφέρατε, περιγράψατε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και τη συζήτηση για την ε, συζήτηση στο ε, μεσοδιάστημα της, του πολιετούς προγράμματος υλοποίησης. Πράγματι, οι διαπραγματεύσεις ε, εξελίσσονται σε μια περίοδο σοβαρής κρίσης για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της ε, γνωμοδότησής σας ε, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2009 Εσεί, συνειδητά υποστηρίζετε μια αύξηση του προϋπολογισμού έτσι όπως ε, τη ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια αύξηση γύρω στο 6% ή οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού. Ε, απλοποίηση κανονισμών. Θεωρείται λογικό ε, εν ώψη της ε, αναθεώρησης, τριετούς αναθεώρησης η Κομισιόν δεν έκανε μια πλήρη αναθεώρηση των κανονισμών, των δημοσιονομικών κανονισμών. Ο κύριος Ιβαν. Καλδίρα pentru acest raport, dar în al doilea rând aș vrea să ridic un semn de întrebare asupra celor 95% de procente a plăților care nu sunt afectate de Δεν έχουμε μετάφραση από τα ρουμανικά, επισημαίνει κάποιος. Α, ούτε και στα δανέζικα. Άρα δεν είμαστε μόνοι, αισθάνομαι καλύτερα τώρα, λέει ο μιλητής. Ωραία, είναι ευχάριστο που δεν είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, Πρέπει να μεταφράσω τα όσα έχω γράψει στα ρουμανικά τώρα για να τα πω αγγλικά. Δεν συμφωνώ με τα όσα είπε ο Επίτροπος Σεμέτα ότι το 95% των πληρωμών ε, είναι απειλαγμένα σφαλμάτων. Ε, και δεν συμφωνώ επειδή γνωρίζω την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μου. Και ο καθένας γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στη δική του χώρα. Και συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολλά λάθη στην ε, χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και υπάρχουν προβλήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αναφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις εθνικές αρχές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι εδώ υπάρχει κενό επικοινωνίας, έλλειψη επικοινωνίας στην ε, διαδρομή δηλαδή από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό. Γνωρίζω την περίπτωση που επικρατεί στη Ρουμανία. Είμαι βέβαιος ότι όταν επισημένονται λάθη ή σφάλματα σε εθνικό επίπεδο δεν κοινοποιούνται ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θεωρώ ότι το 95% είναι, πολύ, ε, είναι μια αισιόδοξη τιμή, αλλά δεν είναι ρεαλιστική. Ως εκπρόσωπος των φορολογουμένων της χώρας μου, θέτω το ερώτημα για τον κανόνα του 50-50 σχετικά με την επιβολή κυρώσεων. Και δεν συμφωνώ ότι τα κράτη θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά τα κονδύλια. Διότι ε, έχουμε περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος είναι επίσης το κράτος, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει δύο φορές, να καταβάλει διπλά ε, για, για ποσά ή για κονδύλια τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ορθώς για κονδύλια δηλαδή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Και το ερώτημα είναι πόσο αξιόπιστες είναι οι εκθέσεις οι οποίες έρχονται από τις εθνικές αρχές και αν το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει, ελέγχει την αξιοπιστία αυτών των εκθέσεων που προέρχονται από τις εθνικές χώρες. Ευχαριστώ, συνάδελφος Μαγιέρ. Κύριε Μαγιέρ, Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό ελεγκτικό Συνέδριο για την έκθεση αυτή που μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα και μέσω των σφαλμάτων ε, που ανέφερε ήδη και ο κύριος ε, Χατζημαρκάκης ε, σφάλματα ιδίω στον τομέα της συνοχής αλλά πάντως εκτός από τους τομείς που αναφέρθηκα νομίζω ότι γενικότερα υπάρχουν λιγότερα σφάλματα θα ήθελα να κάνω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχήν για το θέμα της ε, απλούστευσης. Δεν ε, είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορώ να έχω μακρά εμπειρία. Ξέρω ότι συχνά μιλάμε για τις συνέπειες μεμονωμένων πρωτοβουλειών ε, και εδώ θα ήθελα ε, να μιλήσω ιδιαίτερα για τον τομέα της γεωργίας. Στον τομέα της γεωργίας μπορεί να είναι θαυμάσιο το να έχουμε συστήματα GPS που ελέγχουν αν τα δάση τα οποία έχουν δηλωθεί όντως υπάρχουν, αν οι εκτάσεις που δηλώνονται ότι καλλιεργούνται όντως καλλιεργούνται κλπ. δεν μετρούνται στην πράξη οι επιφάνειες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν ε, πάει κανείς να μετρήσει επιτόπου τέσσερα τετραγωνικά μέτρα στη γωνία ε, της γεωργικής εκμετάλλευσης. Το σύστημα GPS δεν συμπίπτει επακριβώς με το σύστημα μετρήσεων επιτόπου. Μπορεί να μην ε, πρόκειται λοιπόν για απάτη από την πλευρά του Γιώργου που δηλώνει κάτι, αλλά μπορεί με το σύστημα ε, όπως ισχύει, αυτό το οποίο έχει δηλωθεί να ε, φαίνεται ως παρατυπία. Και μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις και πληρωμές που δεν αναλογούν ε, στην πραγματικότητα και μερικές φορές καταποκοπή αναφέρονται ε, κάποια, κάποιες εκτάσεις και γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή να μην οδηγήσει η διαδικασία διόρθωσης ε, σε κυρώσεις εις βάρος των αγροτών που δεν ευθύνονται και σε πολλές χώρες όπως οι σκανδιναβικές χώρες και η Αυστρία και η Γερμανία γνωρίζουν αυτά τα προβλήματα των μετρήσεων ε, και ε, των υπολογισμών μέσω ε, GPS και θέλουμε να φροντίσουμε να εκλείψουν αυτά τα λάθη στο, στο μέτρο του δυνατού. και σίγουρα να αποφεύγονται περιπτώσεις που εκ προθέσεως θα δηλώσει κάποιος κάτι και θα υποφεληθεί από το σύστημα μετρήσεων που εφαρμόζεται μέσω του GPS. Ε, καταλαβαίνετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλοι οι αγρότες θα είναι δυσαρεστημένοι αν πέντε χρόνια αργότερα ανακαλυφθεί ότι οι εκτάσεις που είχαν υπολογιστεί δεν είχαν υπολογιστεί σωστά. Νομίζω ότι είναι να τροποποιηθεί το σύστημα των καταποκοπή υπολογισμών ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο δίκαιο. Ένα άλλο σημείο το οποίο, για το οποίο άκουσα τον κύριο Σέμετα. Ε, γίνεται έλεγχο των διαφόρων χωρών διαφορετικά και με διαφορετικά standards, κάτι το οποίο είναι προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Δεν εξετάζουμε ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμόσει χώρες μεμονωμένα και μπορεί να οδηγηθούμε ε, σε καταστάσεις όπου, παίρνω ένα παράδειγμα από τη δική μου χώρα, μπορεί ε, στη Γερμανία να υπάρχει ε, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να επιδοτηθεί είτε από ε, γεωργικό, γεωργικό προϋπολογισμό είτε από κάποιο κονδύλι για πολιτιστικά θέματα και αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει σε άλλες χώρες γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα προστασίας της φύσης και επειδή δεν υπάρχει αυτό σε άλλα κράτη-μέλη, μπορεί να αξιολογηθεί ως σφάλμα ή ως εσφαλμένη καταβολή χρημάτων και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την εφαρμογή ίδιων διατάξεων ε, ούτως ώστε να μην εμφανίζονται ως ε, σφάλματα ε, κάποιες διατάξεις που υπάρχουν σε μεμονωμένες χώρες και δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Τώρα όσον αφορά την αποστολή περισσότερων ελεγκτών, ίσως να χρειάζεται η αποστολή περισσότερων ελεγκτών στις χώρες όπου υπάρχουν μεγάλες ατασταλίες η γεωργία στη δανία παραδείγματος χάρη έχει ένα θαυμάσιο σύστημα ελέγχου δεν έχει νόημα το σφάλμα του 0,08 να το κατεβάσουμε στο 0,04 θα ήταν περιττό να στείλουμε περισσότερους ελεγκτές σε μια χώρα που η μείωση του σφάλματος δεν μας ωφελεί πολύ. Αν μπορούμε να μειώσουμε όμως το σφάλμα από το 25% στο 20% αυτό θα ήταν πολύ πιο σημαντικό. αν στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα σύστημα GPS ή δεν εφαρμόζεται σωστά είναι προτιμότερο ε, να εντείνουμε τους ελέγχους εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο μείωσης. Να μην προσπαθήσουμε δηλαδή να στείλουμε ελεγκτές στη Δανία να το κάνουμε από 0,5-0,49 αλλά να, το στείλουμε, να το στείλουμε εκεί όπου θα ανταποκρίνεται στην ε, δαπάνη την οποία κάνουμε. Τα ε, χρήματα που δαπανούμε θέλουμε να να είναι προς όφελος των αγροτών και προς όφελος των φορολογουμένων και προς όφελος όφελος των χωρών. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους, θέλουμε να βοηθήσουμε ε, τους ε, πολίτες. Ε, αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Ένα τελευταίο σημείο τώρα. με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να υπάρχει μια ισότιμη εφαρμογή από την πλευρά της Επιτροπής και ισότιμη εφαρμογή σημαίνει ότι ε, δεν θα γίνεται υλοποίηση σε μεγάλο βαθμό από τους μεν, σε μικρό βαθμό από τους δε. Κάτι τέτοιο θα ήταν ε, πηγή προβλημάτων και ε, βλέπουμε πολλές φορές ότι τα ποσοστά υλοποίησης ε, διαφέρουν κατά πολύ και αυτό θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ναι, αλλά θέλω να πω τη γνώμη μου για τους ετήσιους λογαριασμούς, Πρόεδρε. Γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Ο Πρόεδρος διακόπτει. Αγαπητοί συνάδελφε, μπορούμε να έχουμε το λόγο και μισή ώρα, αλλά δεν είναι αυτό που βοηθάει. Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ το λόγο συχνά, αλλά όταν θέλω κάποια στιγμή να εκφράσω τη γνώμη μου για ένα συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι έχουμε το χρόνο και θα πρέπει να μπορούμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας στην Επιτροπή στην οποία βρισκόμαστε για μια δεδομένη, χρον... για μια δεδομένη έκθεση. Αν με διακόπτετε κάθε φορά θα χρειάζομαι ακόμη περισσότερο χρόνο, Πρόεδρε. die Ισότιμη υλοποίηση λοιπόν ήταν το σημείο στο οποίο αναφερόμουν πριν διακόψετε. Θα είχα τελειώσει άμα δεν με είχατε διακόψει. Είναι πολύ σημαντικό σημείο λοιπόν η ισότιμη υλοποίηση και νομίζω ότι εδώ η Επιτροπή πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία και ευχαριστώ για άλλη μια φορά το ελεγκτικό συνέδριο για την παρουσίασή του. Κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρος, πρόθεσή μου δεν ήταν να σας διακόψω, αλλά επειδή όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρέμβουν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι, γιατί 11 και 4, 11 και μισή το αργότερο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Όλα αυτά που λέτε είναι πολύ χρήσιμα στη συζήτησή μας, αλλά από την άλλη θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλου του συναδέρφου να πάρουν το λόγο εξίσου. Δεν μπορεί ο ένα να μιλάει μισή ώρα και άλλο ένα λεπτό. Η συναδέρφο Ιβάνοβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να πω στο Ρουμάνο συνάδελφο ότι ούτε βουλγαρικά υπάρχουν. Δεν είσαστε μόνος δηλαδή χωρίς ε, διερμηνία. Θα μιλήσω λοιπόν αγγλικά. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ το ελεγκτικό συνέδριο για τη δουλειά του. Το είπαν κι άλλοι συνάδελφοι, αλλά κι εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι που βλέπω κάποια πρόοδο σε μερικούς τομείς όπως είναι το Ταμείο Συνοχής. Βέβαια, κατά πόσο θα συνεχιστούν ή όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και στον τομέα της γεωργίας, της έρευνας, της ενέργειας, των μεταφορών, της ε, διεύρυνσης. Πρέπει επίσης να δούμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την ποιότητα των δαπανών. Πώς μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν αυτή η αποτελεσματικότητα. Το θέμα δεν είναι να έχουμε περισσότερους ελέγχους, αλλά να έχουμε περισσότερο αποτελεσματικούς ελέγχους. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται επικοδομητική δουλειά. Εμείς ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε πρόοδο, όπως λέει και ο κύριος Σόντεγκαρτ. Εμείς θέλουμε να διαπιστωθεί πρόοδο σε όλους τους τομεί όπου δαπανώνται χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Ο κύριος Φίλωμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι και σύντομο και προσεκτικός. Δεν είχαμε χρόνο να κοιτάξουμε όλο το υλικό και έτσι δεν μπορώ να αποφανθώ τώρα. Μπορεί να φαίνεται λοιπόν κάπως πρόημο αυτό που θα πω. Αλλά καταρχήν το προφανές. Μπορεί να φαίνεται η τάση θετική, αλλά και εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας ακόμα, κάθε άλλο. Σε μερικούς τομείς μας περιμένουν μεγάλες προκλήσεις που θα ήθελα να τις μελετήσουμε πιο προσεκτικά, όπως είναι η Γεωργία. Εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα και προβλήματα αυξανόμενα. Μπορεί να είναι σύμπτωση βέβαια. Το ίδιο πρέπει να πω και για την Αλία. Αν δείτε τι λέει στην Αλία, σας πιάνει πονοκέφαλος. Αλλά τι, πρόκειται για στατιστική ψευδέστηση ή πρόκειται για κάτι πραγματικό. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Αλλά και εκεί που υπάρχουν ε, βελτιώσεις, στη συνοχή. Από 11 σε 3% πάμε. Ωραία. Αλλά δεν χαιρόμαστε όλοι. Γιατί. Γιατί ε, μας μπαίνουν και ψηλή στα αυτιά. Πρόκειται για σύμπτωση, πρόκειται για φάτα μοργάνα ή πρόκειται για πραγματικές προκλήσεις. Δεν ξέρω. Είναι σαν να έχουμε ένα διάγραμμα που ανεβοκατεβαίνει η γραμμή. Πρόκειται για συμπτώσεις μήπως και τίποτα άλλο. Άκουσα το κύριο Χατζημαρκάκη και τις κυρώσεις. Μα τελικά κουράζεται κανείς να επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια. Είναι πάντα ίδιες χώρες και τα ίδια προβλήματα. Ξανά και ξανά. Και έτσι σκέφτομαι κι εγώ, ωραία τι θα κάνουμε με κυρώσεις. Χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τις κυρώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αν όχι, ας επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό φέτος αν πιστεύουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε τις κυρώσεις που προβλέπονται αποτελεσματικά. Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό που ακούστηκε για τη σύνδεση όλων αυτών με τον προπολογισμό. Γιατί τουλάχιστον για μένα βλέπετε το θέμα των καλών ελέγχων πρέπει να επηρεάζει και τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Αν δεν χρησιμοποιείτε σωστά τις κυρώσεις, τότε... Ε, ωραία, ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για να τις χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της απαλλαγής, να το δούμε αυτό. Μήπως γίνεται. πέρα από το ότι μήπως έχουμε πραγματικά προβλήματα στη γεωργία, στην αλία, στη συνοχή. Εντάξει, αλλά πέρα από αυτό να συζητήσουμε και τι κυρώσεις προβλέπονται και πώς αυτές εφαρμόζονται. Ευχαριστούμε. Ο κύριος για το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα Χωρί να μακρηγορήσω, να δώσω ένα σύντομο παράδειγμα και να μιλήσω για το Ταμείο Συνοχή. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καλτέρα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση ε, τη έκθεση, γιατί η έκθεση του ετήσιου λογαριασμού για μα είναι ένα σημαντικό ε, σημείο προσανατολισμού. βλέπω την πολιτική συνοχής που μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ασθενεί σοβαρά. Ασθενεί από τα περασμένα έτη και βλέπουμε ότι δεν έχει θεραπευθεί ο ασθενή και υπάρχει και κίνδυνο υποτροπής μάλιστα. Και σαφώς ε, καθήκον όλων μας και της Επιτροπής μας είναι ο έλεγχος ε, των δαπανών και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και το θέμα της απλούστευσης παρότι δεν με ακούει η συνάδελφος Χολμάγερ γιατί δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το θέμα της απλούστευσης. τα δύο τρίτα των σφαλμάτων προκύπτουν διότι δεν λειτουργούν σωστά τα συστήματα κρατικών προμηθειών. Όταν ήμουν σε κάποια δημόσια υπηρεσία, θυμάμαι ότι ασχολούμαι με κάποια θέματα κρατικών συμβάσεων, για κάποια θέματα δημοσίων σχέσεων. Και θυμάμαι την όλη διαδικασία που έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Είναι τεράστιος ο όγκος της δουλειάς και πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν θέλουμε να αποφύγουμε σφάλματα. Αυτό είναι το μέλημα όλων μας, αυτό συζητάμε και νομίζω ότι αυτό θα ήταν πρώτη προτεραιότητα. Για το ρόλο των κρατών μελών πρέπει να πούμε ότι ξέρουμε ότι το 80% των χρημάτων τα διατηρίζονται τα κράτη-μέλη και ξέρουμε ότι κατά τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων συμβαίνουν τα σφάλματα και γνωρίζουμε ότι πρέπει να συζητηθεί με τα κράτη-μέλη το πώς θα μειωθεί το ποσοστό σφάλματος στη διαχείριση αυτή. Κανείς δεν ε, είναι άμυρος ε, λαθών και ε, σαφώς το σύστημα ελέγχου δεν είναι πάντοτε απόλυτα αποτελεσματικό και ο Επίτροπος κ. Σέμετα είπε ότι λειτουργεί το σύστημα αυτό με την επικύρωση της Επιτροπής και αυτό ε, το βλέπουμε και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ξέρουμε ότι γίνεται με δειγματοληπτικό έλεγχο και σε σημεία στα οποία έχουν γίνει δειγματοληπτικοί έλεγχοι πολλέ φορέ ε, το ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και πρέπει ε, να εμβαθύνουμε τον έλεγχο των συστημάτων στα κράτη-μέλη. Εδώ υπάρχει ε, λοιπόν το καθήκον των διοικήσεων για ίσπραξη των ασφαλμένων των αχρησίτως καταβληθέντων χρημάτων. Θα ήθελα να πω ακόμη κάτι. Πιστεύω ότι θα πρέπει το θέμα της διεύρυνσης του προϋπολογισμού ε, να συζητηθεί στο κατάλληλο βήμα και δεν είναι ένα θέμα το οποίο ε, είναι προς ε, συζήτηση από τα μέσα ενημέρωσης και από τους δημοσιογράφους. Ε, εμάς μας ενδιαφέρει το να φτάνουν τα χρήματα σε αυτούς στους οποίους πρέπει να φτάσουν, ούτως ώστε να αναπτυχθούν οι πολιτικές τις οποίες έχουμε εγκρίνει και συμφωνήσει. θα μου πείτε ότι ε, στο ποδήλατο χρειάζονται δύο ρόδες και δεν μπορούμε με τη μία ρόδα μόνο να πηγαίνουμε και χρειάζεται ε, η συνεργασία και με την Επιτροπή ε, προπολογισμών για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετούμε τους φορολογουμένους βάσει αυτών τα οποία υπάρχουν στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Γκέρπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Καλντέρα για την έκθεσή του για το έτος 2009. Με μια ε, γρήγορη ανάγνωση και ιδιαίτερα ανάγνωση της σύνοψης θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο να την αναγνώσει κανείς σε σχέση με πέρσι. Αυτό που δεν είδα ακόμα είναι μια γενική περιγραφή των ανομαλιών. Πέρσι ξέραμε ότι είχαμε 11% τέτοια σφάλματα ως προς την συνοχή. Αυτό το κεφάλαιο δεν το βρήκα ακόμα. Ίσως ενδεχομένως μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες από αυτού. Επιπλέον, βλέπω ότι εστιάζεται περισσότερο την προσοχή σας σε σχέση με πέρσι στα συστήματα ελέγχου έναντι του πραγματικού αποτελέσματος του έργου σας. Παρά τα αυτά θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό το ότι σχεδόν σε όλους τους τομείς δεν υπάρχει ένα ικανοποιητικό σύστημα. Και αν κανείς κοιτάξει τις ανομαλίες, αν δεν υπάρχει σύστημα, είναι πολύ δύσκολο να επισημάνει κανείς και να εντοπίσει τις ανομαλίες και να έχει τα σωστά νούμερα. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο σύνθετο χαρακτήρα των κανόνων, με μεγαλύτερη ένταση. Ε, τώρα ασχολούμαστε με το νέο δημοσιονομικό κανονισμό και αυτό είναι σημαντικό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πολλές από τις παρατυπίες οφείλονται ακριβώς στο σύνθετο χαρακτήρα των κανόνων και όχι επειδή κάποιοι θέλουν να παρακάψουν τους κανόνες. Έχω κάποιες απορίες σχετικά με την Γεωργία. Πέρσι είχαμε πράσινο φως στη Γεωργία. Φέτος και πάλι είναι πορτοκαλί το φως. Πέρσι είχαμε πράσινο στη Γεωργία, πράσινο φως, αλλά ε, το, ο τομέας της ανάπτυξης της υπαίθρου ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Μπορείτε να σχολιάσετε την ανάπτυξη της υπαίθρου φέτος. Τώρα, θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα σχετικά με τα, τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια. Άκουσα ότι κάποια ελεγκτικά συνέδρια εθνικά δεν ε, βοήθησαν πάρα πολύ το έργο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έτσι περαιτέρω αυτή τη δήλωση. Ο συνάδελφος Στάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τον κύριο Ιβαν και την κυρία Λανόβα. Δεν υπάρχει και Ολλανδική μετάφραση. Κύριε Καλτέρα, πολλές θερμές ευχαριστίες προς εσάς και τους συναδέλφους σας για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να ε, τη μελετήσουμε, αλλά ρίχνοντας μια ματιά διαπιστώνει κανείς ότι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε είναι το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια. Για μία ακόμα φορά αναφέρεται δύο σημαντικά και πολύ σοβαρά δεδομένα. Στις σελίδες 11 και 12, το επισήμανε και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Πρώτον, οι πληρωμές σχετικά με τους λογαριασμούς του 2009 στη Γεωργία, τη συνοχή, την έρευνα, την ενέργεια, τις μεταφορές, εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη, διεύρυνση, ε, εκπαίδευση, ε, παρουσιάζουν σοβαρούς σοβαρά σφάλματα. Από την άλλη, λέτε ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου είναι εν μέρη αποτελεσματικά ως προς την ανείχνευση, τον εντοπισμό και την διόρθωση ε, πληρωμών. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το μήνυμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Και βεβαίως λέτε ότι φέτος στον τομέα της γεωργίας έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ή ότι υπάρχει μια υποχώρηση σε άλλους τομείς και στη συνοχή είπατε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το βασικό μήνυμα παραμένει το ίδιο. Και το βασικό μήνυμα είναι ότι υπάρχει ένα θεμελιώδες, ένα βασικό πρόβλημα ότι οι χώρες μέλη δεν κάνουν αυτό που όφυλαν να κάνουν και η Επιτροπή τις αφήνει να ξεφεύγουν. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Και η Κομισιόν θα πρέπει να εποπτεύει εάν οι εθνικές αρχές πράττουν αυτό που οφείλουν να πράξουν. Παράδειγμα, παράγραφος 435 δείχνει ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά. Παράγραφος 4.35 λέει τουλάχιστον 30% των σφαλμάτων θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να διορθωθούν από τις χώρες μέλη πριν ε, απαιτηθούν δαπάνες από την ε, Επιτροπή. Άρα οι χώρες μέλη ε, σφάλουν Μέχρι πότε θα δεχόμαστε χώρες μέλη να υπονομεύουν την φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πόσο καιρό ακόμα θα δίνουμε απαλλαγή σε μια επιτροπή, σε μια απαλλαγή, σε μια κομισιόν η οποία επί σειράν ετών αναφέρεται από το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν κάνει επαρχής ελέγχους. Και όταν οι εθνικές αρχές θα πρέπει να προβαίνουν σε δηλώσεις διαχείρισης και δεν το κάνουν, δεν το πράττουν, αρνούνται να το πράξουν. Και κύριε Σεμέτα, απευθύνομαι προς εσάς, διότι έχω δύο σχόλια. Ε, είμαι κάπως απογοητευμένος. Αυτή τη στιγμή ε, επανασυντάσσονται οι δημοσιονομικοί κανονισμοί και υπάρχει η πρόταση για αυτές τις δηλώσεις χρηστής διαχείρισης. Αλλά ζητάτε κάτι δηλαδή την δήλωση η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από έναν πολιτικά υπεύθυνο, από έναν υπουργό και όχι από έναν γραφειοκράτη που εκπροσωπεί την ε, χώρα μέλος. Δηλαδή υποχρεώνεται τους αν υποχρεώνεται τους υπουργούς οικονομικών των χωρών μελών να υπογράψουν αυτή τη δήλωση, θα, θα πρόσεχαν κάπως περισσότερο. Ε, άρα λοιπόν αυτές οι δηλώσεις θα πρέπει να υπογράφονται από αυτούς. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το ψήφισμα για την απαλλαγή για το περσινό έτος. Είμαι βέβαιος ότι το έχει υπόψη το εισηγητής και θα ελέγξει αν, αυτά τα, αν τα υπεσχημένα υλοποιήθηκαν. Αλλά σας θέτω ευθέως ένα ερώτημα. Στην παράγραφο 47 της απαλλαγής πέρσι αναφέραμε μία επιστολή, κάναμε μνήα σε μία επιστολή την οποία είχαν υπογράψει η Ολλανδική και η Σουδική κυβέρνηση όπου απαιτεί το καθοδήγηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποιοι πρέπει να είναι οι παράγοντες κλειδί, οι βασικοί παράγοντες της υπογραφής της εθνικής δήλωσης, εθνικής δήλωσης ε, χρηστής διαχείρισης. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς κύριε Επίτροπε είναι εάν ε, καθορίστηκαν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και αν όχι γιατί. Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, αλλά ήθελα να πω ότι ότι ε, ε, ε, έχει μεγάλη σημασία και το θέμα του περιεχομένου της έκθεσης και στα προηγούμενα χρόνια μιλήσαμε για το θέμα των διαρθρωτικών ταμείων. Τώρα απλώς μας λέτε ότι είναι πάνω από 5% το σφάλμα στον τομέα της γεωργίας. Τι σημαίνει πάνω από 5%, 5,1, 5,2. Θα ήθελα τις ποσοστώσεις να τις βλέπουμε κατά τη στοιχεία με αυτά τα οποία είχαμε δει και τα προηγούμενα έτη. Θα μας ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς ε, ε, ε, πώς υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που λείπουν από την έκθεσή μας. Ενδιαφέρει για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να δούμε πόσο έχουμε προχωρήσει. Αναφέρατε και πληροφορίες για το ΡΑΛ, για τα υπόλοιπα προς καθάριση. Έχουμε 177 ε, δισεκατομμύρια για ε, το ΕΡΑΛ. Ε, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό ακριβώς για την υλοποίηση του προπολογισμού. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που επίσης θα θέλαμε να έχουμε και μας λείπει σαν πληροφορία. Επίσης, κάποιο βαθμός σφάλματο ανακράτος μέλος και αναταμείο θα ήταν πολύ χρήσιμο για μα. Δεν τι έχουμε τι πληροφορίε αυτέ προ το παρόν πρέπει να δούμε τις πληροφορίες για να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένη όταν πρέπει να δω 27 εκθέσεις για 27 κρατημέλη για να μπορέσω να βελτιώσω τη δουλειά μου. Ευχαριστώ. Κύριε Σενάουσερ, ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν, αλλά ένα σημείο θα ήθελα κυρίως να αναφέρω όσον αφορά την Επιτροπή Υπάρχουν ε, ε, ε, στοιχεία για διπλές καταβολές κονδυλίων σε πολύ ψηλό ποσοστό. Τι είναι το σφάλμα αυτό. Είναι σφάλμα των υπαλλήλων που δεν το διαπίστωσαν. Είναι σφάλμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το συνολικό ποσό πόσο είναι. Μπορεί να υπάρχουν τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία έχουν συσσωρευτεί και θα θέλαμε να το ξέρουμε. Και ένα τρίτο σημείο όταν μιλάμε για κυρώσεις. Τα χρήματα τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υπαλλήλων ε, επιστρέφονται. Ε, Η κυρία Ευχαριστώ. Έχω μια μικρή παρατήρηση και μια ερώτηση. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχή που έχω στη διάθεσή μου το έγγραφο αυτό, γιατί όταν πρόκειται για διοικητικέ δαπάνε δεν υπάρχει παρά μικρό σφάλμα. Άρα το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύει ότι το σύστημα ελέγχων είναι αποτελεσματικό. Πολύ καλό γιατί συχνά επικρίναμε τα κονδύλια που πάνε στη δίκηση. Ερώτηση τώρα. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ αναρωτιέμαι για το Ταμείο Συνοχής. Θα μπορούσατε να μας δώσετε πιο συγκεκριμένα δεδομένα παρακαλώ γι' αυτό. Γιατί αυτή μια ακούμε ότι Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις στο Ταμείο Συνοχής, σύμφωνοι, αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Το ακούσαμε αυτό και από άλλους συναδέρφους. Θέλω λοιπόν να ξέρω, είναι σύμπτωση το γεγονός ότι υπάρχει μείωση των σφαλμάτων στο Ταμείο Συνοχής ή πιστεύετε ότι έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί καλά και τα κράτη-μέλη έχουν βελτιωθεί. Είναι αυτό ή είναι σύμπτωση. Έχουμε νέου είδους περιοχές, έχουμε νέου είδους προγράμματα. Θέλω να έχω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί από αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα δεν έχω καταλάβει αρκετά. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος του Καλτέρα και η Κομισιόν βέβαια θα πάρει το λόγο. Και είναι αλήθεια ότι για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε πως μερικές χώρες μέλη είναι η τελευταία μαθητή της τάξης, όπως είπε και ο κύριος Χατζιβαρκάκης όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Η Ισπανία, η Ελλάδα, το Ενωμένο Βασίλειο, εν μέρη επίσης. Εγώ θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, οι έλεγχοι γίνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες μέλη? Και τι γίνεται με το επίπεδο ανεξαρτησίας των ελέγχων δίνουμε μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση της απάτης. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε πραγματικά ανεξάρτητα όργανα που κάνουν τους ελέγχους. Τώρα για τον Επίτροπο Σηματάν, όπως είπε και ο συνάδελφος Στάες, καιρός είναι να αναπτύξουμε νέες σημαντικές πρωτοβουλίες στις χώρες εκείνες όπου εδώ και χρόνια δεν ακολουθούν τους κανόνες όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες, για παράδειγμα. Διατυπώνουμε, ε, διαπιστώνουμε συγγνώμη, πολλές παρατυπίες εκεί ή και απάτες σοβαρές. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει λεπτομερή απάντηση για αυτή την προβληματική. Οπότε θα δώσω το λόγο πρώτα στον Επίτροπο μετά και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Καλντέρα για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθηκαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω εδώ ότι η διαδικασία απαλλαγής μόλις ξεκινάει. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τους άλλους επιτρόπους όσον αφορά τα δικά τους χαρτοφυλάκια, τις δαπάνες στα δικά τους χαρτοφυλάκια. Μπορείτε λοιπόν να ρωτήσετε τον κάθε επίτροπο για τη δικιά του αρμοδιότητα. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στα κύρια σημεία που θέσατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Πρώτον, για αυτά που λέει ο εισηγητής και για το θέμα των κυρώσεων. Πρέπει να σας πω πως ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει όλο και πιο αυστηρά το σύστημα κυρώσεων. Και βλέπετε ότι υπάρχει αύξηση στα ποσά που εισπράττονται και στις διορθώσεις, που ανακτούνται δηλαδή και στις διορθώσεις. Για τα διορθωτικά ταμεία είχαμε 11 αποφάσεις για πάυσεις πληρωμών ή για διακοπές πληρωμών σε ειδικέ χώρες. Αλλά και εδώ βλέπετε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν υπάρξει πάυση πληρωμών, υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος, γιατί τότε η εφαρμογή των προγραμμάτων χειροτερεύει. Προσπαθούμε πάντως να εφαρμόσουμε το σύστημα κυρώσεων πιο αποτελεσματικά, πιο αυστηρά. Έπειτα, όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη για την ίσπραξη, πολύ σωστά το εντοπίζει το λεκτικό συνέδριο, με τα προγράμματα που θα έχουμε στο μέλλον, έχουμε ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης για την ανάκτηση ποσών από τα κράτη-μέλη. Οπότε πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση στη αυτή προγραμματική περίοδο και οι πληροφορίες που θα έχουμε από τα κράτη-μέλη για την ανάκτηση των ποσών θα είναι καλύτερης ποιότητας από ό,τι κατά το παρελθόν. Για τον κανόνα του 50-50%. Πρέπει εδώ να διευκρινίσω ότι ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται ως κύρωση μόνο εάν το κράτος μέλος δεν εφαρμόσει τόσα προβλέπονται για την ε, ανάκτηση. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει γίνει. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο το 100% να επιστρέψει, όχι το 50% μόνο. Ο κανόνας αυτός είναι περισσότερο πειθαρχικός παρά έχει να κάνει με ε, τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Όταν μιλάμε τώρα για το 24% στην εκπαίδευση, 62% όπως είπε ο κ. Μπαλσίτης στην οικονομία και τα δημοσιονομικά. Είναι η συχνότητα του λάθους, δεν είναι το επίπεδο του σφάλματος. Στην εκπαίδευση το ποσοστό σφάλματος είναι 2 με 5% όπως είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έρχομαι εδώ τώρα στο θέμα της αποδοτικότητας των ε, δαπανών και της εκθέσεις αξιολόγησης τις οποίες αναφερθήκατε στις παρατηρήσεις σας. Και εγώ περιμένω να δω τις εκθέσεις αυτές, τις αξιολογήσεις αυτές. Είναι σημαντικό να δούμε τους δείκτες αποδοτικότητας και να δούμε σε ποια προγράμματα μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα την απόδοση. Πάντα δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. αλλά πρέπει να το κάνουμε και ορίζοντας τα προγράμματα στη νέα προγραμματική περίοδο. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ, ώστε να υπάρχουν οι προβλέψεις αυτές στους συγκεκριμένους τομείς δαπανών. Για τις απλοποίησεις τώρα. Είναι το θέμα το οποίο έχει τεθεί ξανά και ξανά. Το Δεκέμβριο θα έχουμε μία ανακοίνωση για τις απλοποίησεις όσον αφορά το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η ιδέα είναι να έχουμε μια συστηματική προσέγγιση για τις απλοποίησεις και μια συντονισμένη προσέγγιση Δηλαδή όχι ξεχωριστά κάθε πρόγραμμα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα πλαίσιο για τις απλοποίησεις. Αν κοιτάξετε την ανακοίνωση για την αναθεώρηση του προπολογισμού, θα δείτε την βασική αρχή που διέπει την ανακοίνωση αυτή και που είναι η πρόθεσή μας να έχουμε κανόνες ανατομέα που να συνδέονται άμεσα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται στην νομοθεσία ανατομέα. Και μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη για δικό σε έναν δικό τομέα νομοθεσίας, τότε μπορεί να γίνει κάποια εξαίρεση. Πάντως είναι σημαντικό οι δημοσιονομικοί κανονισμοί να διέπουν τις δαπάνες. όσον αφορά την διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα εδώ είναι η αυστηρή τήρηση των ε, ρυθμίσεων που έχουμε και των κανονισμών μας. Για το 2007-2010, αυτή την προγραμματική περίοδο, τα πράγματα είναι καλά και είναι καλό η εφαρμογή να γίνεται αυστηρά, ο έλεγχος επίσης και να υπάρχουν και κυρώσεις κάθε φορά που ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις απαιτήσει που απορρέουν από την νομοθεσία. Στην πρόταση για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών προτείνονται δηλώσεις εθνικής διαχείρισης που να βελτιώνουν έτσι την απόδοση λογαριασμών των κρατών μελών. Εδώ υπάρχει και το θέμα του κύριου που λέει ποιος τελικά θα, θα υπογράφει τη δήλωση. Η ιδέα μας ήταν αυτή τη δήλωση να την υπογράφει αυτός που είναι στο επίπεδο διαχείρισης και να εφαρμόσετε η ίδια αρχή που έχουμε και εδώ στην Επιτροπή που είναι ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο σκαλοπάτι της διαχείρισης. και εκείνο έχει την ευθύνη της κάθε δαπάνης. Θέλουμε να διατηρηθεί λοιπόν η δήλωση στο κατάλληλο διαχειριστικό επίπεδο κάθε φορά. Τώρα βέβαια στους, για τους δημοσιονομικούς κανονισμούς γίνεται συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, οπότε τελικά εσείς μεταξύ σας θα αποφασίσετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της αναθεώρησης αυτής. Κάποια συγκεκριμένα τώρα ζητήματα που θέσατε. Την κατεύθυνση των δημοσιονομικών δηλώσεων θα είδατε στην ε, ατζέντα μας τι προβλέπουμε για φέτος. Όντως, Είμαστε στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας και θα είμαστε έτοιμοι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Για τις κρατικές προμήθειες τώρα. Ο πρόεδρος Καλτέρα είπε ότι οι κρατικές προμήθειες είναι ένας από τους τομείς όπου έχουμε τα περισσότερα σφάλματα. Συμφωνώ ότι οι κανόνες για τις κρατικές προμήθειες είναι περίπλοκοι και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει κατάρτιση για τους διαχειριστές των ε, ταμείων, των κονδυλίων, όταν πρόκειται για τις κρατικές προμήθειες. Εκδίδουμε και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων στις κρατικές προμήθειες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε και να απλοποιήσουμε κάπως τους κανόνες για τις κρατικές προμήθειες. Αλλά και πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί συλλογικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το σύνολο των Επιτρόπων. Εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες για το 95% δαπανών άνευ σφάλματος. Δεν το εφήβρα εγώ. Χρησιμοποίησαμε τα δεδομένα του ελεγκτικού συνεδρίου και θα δείτε στην έκθεση ότι για πρώτη φορά το επίπεδο σφάλματος ολόκληρου του προπολογισμού είναι της τάξης 2 με 5%. Οπότε αν το κοιτάξετε από την ανάποδη μεριά θα δείτε ότι τουλάχιστον 95% των κονδυλίων είναι άνευ σφάλματος. Είναι μεγάλο επιτεύγμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βοήθησε σίγουρα και το Κοινοβούλιο σε αυτό με, την δικιά του, με το δικό του έλεγχο και με τόσα έγινε κατά τη διαδικασία απαλλαγή. Πάντως, δεν πρέπει να πούμε ότι εδώ τελείωσε η δουλειά μας. Όχι. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Υπάρχουν τομείς όπου μπορεί να γίνει πρόοδος ακόμα. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την κατάσταση όσον αφορά την οικονομική διαχείριση των κοινωτικών κονδυλίων. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στον Πρόεδρο Καλτέρα για τα συμπεράσματα. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα και έχετε στη διάθεσή σας μόνο μισή ώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα καταβάλω προσπάθεια ώστε να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα και τα σχόλια. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας σχόλια και τον κύριο Χατζημαρκάκη και τα μέλη της Επιτροπής. Τα ευχαριστώ θερμά. Το ελεκτικό συνέδριο πράγματι επιδιώκει να προσφέρει σε αυτή την Επιτροπή και σε αυτό το όργανο ε, την βέλτιστη δυνατή έκθεση με πολύ καλό ποιοτικό επίπεδο. Ε, ε, ε, Μας είπατε ότι η παρούσα έκθεση δίνει λιγότερες πληροφορίες σε σχέση με πέρσι. Εκπλήσωμε, διότι κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Προσφέρουμε περισσότερα στοιχεία για κάθε τομέα δείχνουμε ακριβώς ποια είναι τα σημεία ε, σφαλμάτων σε κάθε πολιτική. Και στο τομέα της συνοχής για πρώτη φορά λέμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες. Και ε, το να λέμε ότι πέρσι και πρόπερσι ότι τουλάχιστον το 11% των δαπανών στην ε, συνοχή ε, ήταν ε, εσφαλμένες ενώ φέτος ακριβώς επισημαίνουμε ότι τουλάχιστον το 3% δεν θα έπρεπε να καταβληθούν 3% των πληρωμών δηλαδή και εδώ υπάρχει μια προειδοποίηση δεν θα επαναλάβω τα όσα λέγονται στην έκθεση. Περισσότερες πληροφορίες επί των συστημάτων, πράγματι. Διότι δεν μπορούμε να ε, εξηγήσουμε τα σφάλματα εάν δεν ξέρουμε τα αίτια. Γι' αυτό εστιάζουμε την προσοχή μας στα συστήματα. Η, Έχουμε την, τον ίδιο βαθμό έντασης ως προς ε, την εστίαση και στα συστήματα και στο περιεχόμενο τα προβλήματα, οι αδυνομίες στην διαχείριση και τον έλεγχο οφείλονται στα συστήματα τόσο είτε σε επίπεδο Κομισιόν είτε σε επίπεδο χώρας μέλους. διότι εξακολουθούμε να έχουμε σφάλματα, λάθη. Αυτό είναι σαφές. Και λέμε ότι αν δεν επιληθούν αυτά τα προβλήματα Και ζητώ συγγνώμη που λέω ότι αυτό δεν είναι ούτε σύμπτωση ούτε θαύμα. Αν δεν επιληθούν αυτά τα προβλήματα θα έχουμε την ίδια εικόνα. Για ποιο λόγο ο τομέας της συνοχής έχει τα αποτελέσματα που έχει φέτος. Αν κοιτάξετε την αξιολόγηση 16 επιχειρησιακών προγραμμάτων θα διαπιστώσετε ότι για τις βασικές προδιαγραφές ως προς την ε, διαχειριστική αρχή, την αρχή επιστοποίησης και την αρχή ελέγχου, ο πίνακας είναι σχεδόν πράσινος. Και αυτή είναι μια πολύ σχετική αλλαγή, σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα σημάδι, σήμα ότι το νέο σύστημα για το ε, την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ότι το σύστημα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Είναι αποτελεσματικός προς το κόστος, χρησιμοποιούμε τα κονδύλια. Πρέπει να επισημάνω ότι το ποσοστό υλοποίησης του πακέτου δαπανών στον τομέα της συνοδηγής είναι ενδεχομένως χαμηλότερο. Αν κοιτάξετε τις τιμές υλοποίηση στην έκθεση μας, στο κεφάλαιο της συνοχής, θα διαπιστώσετε ότι οι ενδιάμεσες και οριστικές ε, πληρωμές ε, ισούνται με 23 εκατομμύρια. Αν στο τέλος του 2009 το ποσοστό υλοποίησης ήταν το 1 τέταρτο και είμαστε ήδη στο 2009, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ε, αργή υλοποίηση. Καθυστέρηση δηλαδή. Αλλά όπως ε, λέμε και στον τραπεζικό τομέα, τα κέρδη του παρελθόντος δεν εγγυώνται και τα κέρδη του μέλλοντος. Εδώ υπάρχει μια προειδοποίηση. Πρέπει δηλαδή να διατηρήσουμε τα συστήματα ε, μάλλον να βελτιώσουμε τα συστήματα στο βέλτιστο δυνατό βαθμό. Και αυτό είναι ευθύνη των εθνικών αρχών. Και βεβαίω αυτή τη στιγμή. Ε, αυτή η στιγμή είναι πολύ δύσκολη στιγμή για τι χώρε μέλη, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά στη Γεωργία, να σχολιάσω και αυτό. Τι παρατηρούμε. Για ποιο λόγο τα πράγματα στη Γεωργία είναι διαφορετικά από το παρελθόν. Ακριβώς επειδή τα προβλήματα στο σύστημα παραμένουν. Το Ελεκτικό συνέδριο εδώ και 5-6 χρόνια λέει ότι το βασικό σύστημα διαχείρισης των δαπανών στη Γεωργία ε, πρέπει να εσωματωθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου. Και επί σχεδόν ε, πήρε σχεδόν μια δεκαετία για τις 15 ε, χώρες μέλη και μετά τις νέες χώρες μέλη να ενσωματωθούν. Ε, είχαμε ένα πρόβλημα υλοποίησης με την Ελλάδα και η Κομισιόν και η χώρα μέλος κατέβαλαν προσπάθεια. Τώρα όμως δεν είναι 15 χώρες μέλη, έχουμε 27 χώρες μέλη που πρέπει να εφαρμόσουν το σύστημα και να το διαχειριστούν με επιπλέον νέα μέτρα, πιο επικίνδυνα μέτρα σε σχέση με το παρελθόν. Αν κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση λοιπόν, όπως κάνουμε στην έκθεση, το χρώμα στη Γεωργία είναι πολύ πιο κόκκινο σε σχέση με τη συνοχή. Αν υπάρχουν λοιπόν αδυναμίες στα συστήματα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατυπώσει δύο επιφυλάξει στην ετήσια έκθεση για τη Γεωργία. Η ε, Κομισιόν απαντάει με απόλυτη σαφήνεια στις επιφυλάξεις μας. Έχουμε περισσότερα προβλήματα ως προς την διαχείριση των κονδυλίων στον τομέα της γεωργίας σε σχέση με το παρελθόν. Και πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε αυτό και μετά να απαντήσουμε στο γιατί υπάρχει καθυστέρηση η πιο αργή λειτουργία. Ε, είναι όπως τις ασθένειες ας πούμε. Αν έχει πάθει κάποιος μία λίμωξη δεν μπορεί να την καταπολεμήσει με ασπιρίνη, πρέπει να πάρει αντιβιωτικό. Και έρχομαι και στην κυρία Σόντεγκρατ. Τα σφάλματα δεν είναι πάντα προϊόν απάτης. Ένα σφάλμα ένα λάθος είναι μη συμμόρφωση προς τους κανόνες. Υπάρχει ένα στοιχείο εκεί. Και πρέπει να δούμε αν υπάρχει πρόθεση για την παρέκκληση από τον κανόνα που είναι η απάτη ή όχι. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα σφάλματα που εντοπίζονται μεγάλη τους πλειοψηφία δεν είναι απάτες. Αν υπάρχει έστω και υποψία απάτης, το ελεγκτικό συνέδριο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσει το θέμα στον Όλαφ. Το, οι τρεις περιπτώσεις είναι ένας μέσος όρος. Πολύ περισσότερες περιπτώσεις ε, διαβιβάστηκαν στον Όλαφ, όχι μόνο τρεις. Αν δηλαδή στους ελέγχους που κάνουμε διαπιστωθεί υποψία, υπάρξει υποψία απάτης, γιατί το συνέδριο δεν μπορεί να αποφανθεί αν κάτι, κάποια περίπτωση είναι απάτη ή όχι. Το προωθούμε στον Όλαφ. Δηλαδή αυτό που εμείς αποκαλούμε απάτη δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι μια εκπροθέσεις σφάλμα, συγγνώμη, ε, αυτό που αποκαλούμε σφάλμα δεν είναι μια εκπροθέσεως παρέκκληση ή εκ μη συμμόρφωση προς τον ε, κανόνα. Διάφορα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στο θέμα της απλοποίησης των δημοσιονομικών κανονισμών και για την εφαρμογή ενός συστήματος πιο αποτελεσματικού ως προς το κόστος. Εκεί συνιστώ να κοιτάξετε τη γνωμοδότηση ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Η γνωμοδότηση ε, εστάλει στο σώμα την περασμένη εβδομάδα και με χαρά θα την παρουσιάσουμε όποια στιγμή θέλετε κύριε Πρόεδρε ε, στην Επιτροπή αυτή για να σας αναπτύξουμε τα διάφορα σημεία. Διότι τα, τα προβλήματα ή τα θέματα τα οποία προκύπτουν από τα νέα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου υπάρχουν. Αν θέλουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, αυτή είναι η στιγμή. Τώρα πρέπει να το πράξουμε και έχουμε ήδη εκδώσει τη γνωμοδότησή μας. Θέλουμε να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο διαχείρισης και ακριβώς αυτό το πλαίσιο απαντά στα τέσσερα ερωτήματα. Και τούτο αφορά την περίοδο μετά το 2013. Και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η νομοθεσία ανατομέα και τα διάφορα προγράμματα θα πρέπει να είναι ουσιαστικά το μέσο, το εργαλείο. Διότι πολλά εξαρτώνται από την νομοθεσία κατά τομέα. Η κυρία Αντριάσεν ε, ρώτησε αν υπάρχει μια θετική τάση στην έκθεσή μας. Απάντηση. Παράγραφος 526. Ε, ναι, υπάρχει θετική τάση. στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μέλη και τα θεσμικά μας όργανα λειτουργούν. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αυτή η τάση. Δεν έχει παγιωθεί αν θέλετε και πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά ώστε η κατάσταση να μην ε, ανατραπεί, αναστραφεί στο μέλλον. το ελεκτικό συνέδριο δεν μπορεί να κάνει σχόλια για την διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Εμείς ελέγχουμε την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για τον προϋπολογισμό παρά μόνο εάν ε, τροποποιηθεί η συνθήκη. Ωστόσο οι δημοσιονομικές προοπτικές έχουν πολυετή χαρακτήρα. Και αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μελετήσετε. κάποια μέλη έθεσαν το θέμα της συνεργασίας με τα εθνικά όργανα. Κοιτάξτε, υπάρχει μία ανεξαρτησία από αυτού και ο κύριος Ρεμπαλιά το σχολίασε και ο κύριος Εύαν έθεσε το θέμα των εθνικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Νομίζω ότι έχουμε καλή συνεργασία με τα εθνικά θεσμικά όργανα. Και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο πιλωτικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνεται συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο επί τόπου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία με τα εθνικά το ένα είναι με το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο της Ολλανδίας και το άλλο της Τσεχίας. Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, διότι εδώ εστιάζουμε την προσοχή μας στις αγροτικές δαπάνες. Και αν ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων, θα είναι πολύ ευχάριστο και θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτή η εμπειρία σε ποιο βαθμό αυτή η εμπειρία μπορεί να επεκταθεί και στις άλλες χώρες μέλη. Βεβαίως η συνεργασία εδράζεται στη συνθήκη, στο πνεύμα εμπιστοσύνης και του σεβασμού της ανεξαρτησίας των οργάνων. Πάντα το δηλαδή πρόκειται για μία ε, εθελοντική αν θέλετε συμμετοχή από πλευράς των χωρών μελών. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και ελπίζουμε να υπάρχει το ίδιο ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας και από την άλλη πλευρά. Τα εθνικά θεσμικά όργανα είναι ανεξάρτητα, όπως σας είπα. Πέρσι, όταν είχαμε τη συνάντηση με τους 27 επικεφαλείς των εθνικών οργάνων, διατυπώθηκαν κάποιες ανησυχίες ως προς την ανεξαρτησία των εθνικών ελεγκτικών οργάνων. Υπάρχουν Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποια περιφερειακά όργανα και στείλαμε μια επιστολή Α, επισύροντας την προσοχή υποψηφίων ε, χωρών, ε, όχι χωρών μελών, ε, στο ζήτημα αυτό της ανεξαρτησίας των εθνικών ελεγκτικών οργάνων. Ένα θέμα είναι η ανεξαρτησία των εθνικών φορέων που είναι επιφορτισμένα για την σύνταξη των εκθέσεων και εσείς κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε σε αυτό όταν θέσατε το θέμα εκεί το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει την ευθύνη να αξιολογήσει την ανεξαρτησία αυτών των θεσμικών οργάνων. Υπάρχει βεβαίως η απέτηση της ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και στο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο υπάρχουν, υπάρχουν ε, τέτοιες δικλείδες ασφαλείας και από πλευρά εθνικών αρχών ως προς τον τομέα της γεωργίας παραδείγματος χάρη. Εκεί δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση της ανεξαρτησίας. Εμείς αξιολογούμε τις επιδόσεις αυτών των ε, θεσμικών οργάνων και τα συστήματα αναφοράς. Και βεβαίως οι εκθέσεις αυτές απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι στο ελεκτικό συνέδριο. Και εμείς επίσης αξιολογούμε τους εσωτερικούς ελέγχους. Δηλαδή ελέγχουμε και τα συστήματα και αναφέρουμε, κοιτάζουμε το, στο έργο, κοιτάζουμε το έργο αυτών των οργάνων και το αποτέλεσμα των, της δράσης τους. Και αξιολογούμε αυτό το έργο στο πλαίσιο της εποπτικής ευθύνης που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο ερώτημα από τον κύριο Γκρέσλερ. για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια δήλωση διασφάλισης. Μια δήλωση αξιοπιστίας ανά χώρα μέλος. Καταρχήν η συνθήκη δεν το επιτρέπει και δεύτερον δεν θα ήταν ε, αξιόπιστο κάτι τέτοιο, διότι δεν διαθέτουμε όλα τα μέσα, όλους τους πόρους. Το επεσήμανε και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Η Κομισιόν θα πρέπει να μας δίνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία επί τη βάση των ελέγχων που αυτή κάνει. Εμείς ως εξωτερικός φορέας ελέγχου αξιολογούμε την αξιοπιστία των διαβεβαιώσεων που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι υπάρχει το εσωτερικό σύστημα ελέγχου που βασίζεται στο έργο των χαμηλότερων επιπέδων. Η το να, το οικοδομεί κανείς δηλαδή τον εσωτερικό έλεγχο επί τη βάση ελέγχων που γίνονται σε χαμηλότερο επίπεδο, επίπεδο είναι φυσιολογικό και μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εποπτεύουσα αρχή μπορεί να μας δώσει τις πληροφορίες που εμείς θέλουμε. Και βεβαίως εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε αν τα στοιχεία που μας δίδονται είναι αξιόπιστα ή μη αξιόπιστα. Σχετικά με τις ε, ε, ε, κρεμούσες υποχρεώσεις στον τομέα της συνοχής και την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανακεφάλαιο. Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες ως προς τις υποχρεώσεις των τομέα της συνοχής. Σελίδα 149 του προϋπολογισμού. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του αριθμού των εκκρεμουσών υποχρεώσεων στις πολιτικές της συνοχής, κοινωνική πολιτική κλπ. Όπως το επεσήμανε και ο Επίτροπος ε, Σεμέτα. Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι αυτό το όργανο που ξεκινά τώρα την διαδικασία της απαλλαγής και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε απόλυτα στην, όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε τη βούληση να συνεργαστούμε και να σας βοηθήσουμε. Αν υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία, στα οποία δεν απήντησα, με χαρά θα απαντήσω γραπτός, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και θεωρώ ότι είναι η στιγμή να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το ζήτημα της αναθεώρησης, της μεταρρύθμισης. Μοναδική ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γνώμη του ελεγκτικού συνεδρίου ε, πάνω στην, ε, στο αναθεωρημένο στους αναθεωρημένους δημοσιονομικούς ε, κανονισμούς. Και αυτό θα το πράξουμε με απόλυτη ευθύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντησή σας. Και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χατζημαρκάκη. Ξέρω ότι βιάζεται ο πρόεδρο να φύγει και δεν θα καθυστερήσω. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είμαι ευγνώμων προ τον κύριο Σέμετο τον Επίτροπο, για τον πολύ ανοιχτό χαρακτήρα και για αυτά τα οποία μα είπε, για τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή βάση για πολύ επικοδομητική συνεργασία μας με την Επιτροπή. Όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία που κάπως συγκεκαλυμμένα εμφανίζονται στην έκθεση και δεν ε, φαίνονται τόσο ξεκάθαρα, όντως ε, η έκθεση αυτή ε, είναι κάπως είναι σαν να συγκαλύπτει κάπως τα στοιχεία. Βλέπουμε το 3%, αλλά το 3% δεν λέγεται ότι είναι αυτό το οποίο δεν έπρεπε να έχει καταβληθεί. Ε, θα έλεγα ότι είναι κάπως κωδικοποιημένα και πρέπει να ψάξει κανείς να τα βρει τα στοιχεία. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια ε, παρεξήγηση στο, όσον αφορά την κοινή γνώμη. Και η κυρία Χολμάγερ επίσης τόνισε αυτό το σημείο και είναι σημαντικό να τονίζουμε το τι σημαίνει σφάλμα. Υπάρχουν σφάλματα τα οποία ε, δεν γίνονται εκ και σφάλματα τα οποία γίνονται εκ όταν μιλάμε για την απλούστευση πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να εμβαθύνουμε και συμφωνώ με τον ε, Επίτροπο. Είμαι ευγνώμων που είπατε ότι θα πρέπει σε κεντρικό επίπεδο να ασχοληθείτε με την ε, απλούστευση. Όντω, σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να ξεκινήσει η απλούστευση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Καλντέιρα, για την έκθεση αυτή, διότι βεβαίω και υπάρχει μια θετική τάση συνολικά, αλλά αναφέρονται τα σφάλματα συγκεκριμένα και ακριβώς μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τις τάσεις που υπάρχουν. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέντευξη τύπου στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που απίθυναν και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. Καλτέρα και τον Επίτροπο κ. Σεμέτα.